Uh, so good morning, everybody. I think we can make a start. If everyone would like to take their places. Um, and, uh... Καλημέρα σας. Παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε. Έχουμε πολύ φορτωμένες ε, συνεδρίες, τρεις στον αριθμό. Να σας καλωσορίσω όλους. Να επιβεβαιώσω την ημερήσια διάταξη για την, επόλυπη, την επόμενη μία μισή μέρα. Μία αλλαγή έχουμε μόνο για τη γνωμοδότηση για τις διατραπεζικές προμήθειες θα την εξετάσουμε αύριο το πρωί μετά τις ψηφοφορίες. Να σας υπενθυμίσω ότι θα αρχίσουμε στις 9 και 4 αύριο. 9 και 4 για να μπορούν να συνενώσουν ε, τις ε, δυνάμεις τους ε, οι πολιτικές ομάδες, να τις συγκεντρώσουν για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε αποτελεσματικά. Ε, τώρα που πλησιάζουμε προς το τέλος της κοινοβουλευτικής ε, θητείας. Οπότε να έχετε τις ομάδες σας έτοιμες για τις 9 και 4 αύριο το πρωί. Καλωσορίζω και τον κόσμο που μας παρακολουθεί από το διαδίκτυο. Ελπίζουμε να μπορέσετε με ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε τις εργασίες μας. Μερικά ακόμα σημεία να αναφέρω. Είμαστε μια πιλωτική επιτροπή για τις ε, συνεδριάσεις ε, χωρίς ε, έγγραφα. Μπορείτε όλα τα έγγραφα να τα λάβετε στους φορητούς υπολογιστές σας ή στις πινακίδες αφής σας. Θα γνωρίζετε ότι είναι Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Ομάδα που είναι γύρω από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, αφορά κυρίως ε, οικονομικές ε, εκθέσεις και εκθέσεις απασχόλησης. Ε, είναι κάτι για το οποίο βέβαια δεν έχουμε προετοιμαστεί εγκαίρως στη σημερινή μας συνεδρίαση. θα θέλαμε να συμμετέχουμε περισσότερο στην κοινοβουλευτική ομάδα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με ζητήματα εσωτερικής αγοράς και ζητήματα καταναλωτών για την επόμενη χρονιά, εφόσον δεν τα καταφέραμε πολύ καλά φέτος, να σας επιστήσω την προσοχή ότι έχουμε δημοσιεύσει μία έκθεση πλήρη σε πολλές γλώσσες για την πρόσφατη αντιπροσωπεία μας στην Κίνα τέλη Οκτωβρίου. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που αναφέρονται όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων των καταναλωτικών. Επίσης, έχουμε και τα πρακτικά της συνεδρίασης 16ης και 17ης Δεκεμβρίου. Αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις θα θεωρηθούν εγκεκριμένα μέχρι το πέρας της σημερινής συνεδρίασης. Αυτά με τις ανακοινώσεις του Προέδρου. Θα ακούσουμε τώρα ενημέρωση για τους τριμερείς διαλόγους ε, από τα μέλη της Επιτροπής μας που συμμετέχουν σε τριμερείς διαλόγους. Που συμμετέχουν ή θα ήθελα να συμμετέχουν, γιατί δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι τμήμα της διαφάνειάς μας, της προσπάθειας ε, διαφάνειας ε, για διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε πρώτη ανάγνωση. Γιατί ξέρετε ότι είναι εμπιστευτικέ. Α, βλέπω ότι έχω μία φωτογραφία στο ενημερωτικό φυλάδιο αυτού του μηνός. Βλέπω το πρόσωπό μου. Συγγνώμη συνάδελφοι. Α, είναι επειδή σας απίφθηνα ένα μήνυμα με την ευκαιρία της νέας χρονιάς. Με ευχές. Τέλος πάντων το λέω για τους ε, ε, όσους μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο, ότι υπάρχει αυτό το ενημερωτικό φυλάδιο είναι και το προσωπικό της ΣΥΜΚΟ στην πίσω πλευρά του φυλαδίου. Σας εύχονται όλοι καλή χρονιά. Δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και το προσωπικό της γραμματείας. Τέλος πάντων, θα σας το διανύμουμε και αν θέλετε εσείς ε, από το διαδίκτυο να το λάβετε, μπορείτε να μας στείλετε ένα email για να σας το αποστείλουμε ηλεκτρονικώς. Λοιπόν, διαπραγματεύσεις τριμερούς διαλόγου. Η κυρία Κον ε, μετά η κυρία Σαλντεμόσε και μετά η κυρία Πιετικάινεν που περιμένουν ε, να δουν τι θα γίνει με τον τριμερή ε, διάλογο. Θα μας εξηγήσει γιατί. Για τη μεταφορά των, ε, των οχημάτων. Ε, έχουμε τώρα ε, συμφωνήσει ως προς αυτό. Πρώτα η κυρία Κόλιν Λάγκεν να μας πει πού βρισκόμαστε με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχαμε δύο διαπραγματεύσεις, χτες ήταν η τελευταία Νομίζω ότι είναι καλό το πακέτο που καταρτήσαμε. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι η φάση δοκιμής να περιλαμβάνεται, να αποσυνδεθεί η προθεσμία για τα πρότυπα και ε, την εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Αυτό ήταν ε, απέτηση του Συμβουλίου για να ε, βοηθηθούν τα κράτη-μέλη κατά την εφαρμογή. Ένα πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, οι προθεσμίες για την εφαρμογή. Ίσως θα το θυμάστε και εδώ στην ΙΜΚΟ είχαμε μια μεγάλη συζήτηση. Ήταν 48 μήνες η προθεσμία του Αντρέα Σουάμπη πρόταση, μέχρι 15 μήνες από τον κύριο Χρόιτσμαν και τον κύριο Ταραμπέλα. Είχαμε 15 μήνες και για την κεντρική αρχή και μια διαφορετική για την υποκεντρική, 30 δηλαδή. 36 είχαν προτείνει για την τα υποκεντρικά. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, υπερβολικά μεγάλο. το Συμβούλιο είπε 24 και 30 αντίστοιχα μήνες και αυτό πιστεύουμε ότι είναι πολύ μεγάλο διάστημα ε, δεδομένων των μεγάλων ελαφρύνσεων που πετύχαμε για την εφαρμογή. Πιέσαμε να προσθέσουμε δύο αιτιολογικές σκέψεις για να υποχρεώνεται η Κομισιόν να ε, παράσχει την απαραίτητη βοήθεια. Σε αυτό το σημείο το Συμβούλιο, το οποίο το κατάλαβε χθες, το θέμα πως έχει και μας υποσχέθηκε ρητά ότι θα έρθει την Παρασκευή. Ο πρόεδρος ε, απίφθινε επιστολή και στους μόνιμους αντιπροσώπους της Ελλάδας και φαίνεται ότι θα περάσουν οι πιο μικρές προθεσμίες. Αλλιώς και το χρονικό διάστημα εφαρμογής θα είναι υπερβολικά μεγάλο. Εμείς τώρα έχουμε φτιάξει ένα μεγάλο πακέτο με τις αναθέσεις, με την οδηγία για τις ε, παραχωρήσεις, ε, την ανάθεση και ε, το πεδίο εφαρμογής των δύο ετών είχε αναφερθεί εκεί. 36 μήνες μέχρι να καταρτήσει τα πρότυπα η Κομισιόν και 18 για τις ε, κεντρικές ε, και τις 24 για τις ε, μη κεντρικές υπηρεσίες ανάθεσης. Αυτό είναι καλό. Δουλέψαμε κάτω από χρονικές πιέσεις. Πολλές φορές δουλέψαμε μέχρι αργά τη νύχτα. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τους κοιόδης εισηγητές για τη βοήθειά τους. Ήταν πολύ καλή η συνεργασία και χθε ο Πρόεδρος άσκησε μεγάλη επιρροή στο Συμβούλιο για να ανταποκριθεί στο αίτημά μας για τις προθεσμίες. Συνολικά καλό το αποτέλεσμα, πολύ καλό. Ευχαριστώ. Υπογραμμίζω και εγώ, όπως είπες και εσύ στην αρχή, ότι αυτό είναι ένα πακέτο το οποίο συμφώνησε να το βάλει η Ελληνική Προεδρία στην Κορεπέρ, την Παρασκευή, δεν έχουμε τελειώσει δηλαδή. Ο Έλλην Πρόεδρος ε, θα υποστηρίξει, θα υποστηριχθεί. Έστειλα επιστολή στον πρόεδρο της Ελληνικής Προεδρίας εγκρίνοντας την προσέγγιση που υιοθετήσαμε. Να ευχαριστήσουμε και την Κομισιόν όμως που έκανε δημιουργικές και επικοδομητικές προτάσεις και για τις παραχωρήσεις και <clears throat> την πειθό στα κράτη-μέλη για να προχωρήσουν το θέμα. Ελπίζομαι λοιπόν την επόμενη εβδομάδα να επισημοποιηθούν τα αποτελέσματα. Αν είστε σε επαφή με τις κυβερνήσεις σας πάνω σε αυτό το θέμα, θα βοηθήσει να πείτε μια καλή κουβέντα για τη συμβαστική λύση. Για την ε, εποπτεία της αγοράς, ποιος θα παρουσιάσει το θέμα, η Κρίσταλ. Είναι τελείωτη ιστορία αυτό το πακέτο. Και μέχρι τώρα δεν ξεκίνησαμε διαπραγματεύσεις. Όμως Σήμερα η Ελληνική Προεδρία παρουσιάζει πρόταση εντολής στο Συμβούλιο. Και έχουν κάποιο συμβιβασμό. Για το καυτό θέμα του άρθρου 7 δεν ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ελπίζω το καλύτερο δυνατό. Ίσως όμως δεν επαληθευτεί αυτό. Στείλαμε επιστολή στο Συμβούλιο. Εκεί λέμε ότι είναι τεράστια η χρονική πίεση. Άρα τώρα πρέπει να διαπραγματευτούμε. Το στείλαμε το μήνυμα. Ήρθα σε επαφή με τον αρμόδιο Έλληνα Υπουργό και συζήτησα και με άλλα κράτη-μέλη. Όμως άφησα να εννοηθεί ότι πρέπει τώρα να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Αν δεν το κάνουμε αυτό δεν έχουμε χρόνο να διεκπαιρεώσουμε το ζήτημα πριν το τέλος της θητείας. Ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί σήμερα όμως, σχεδιάζουμε ψηφοφορία στην Ολομέλεια όσον αφορά την έκθεση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη το κίνδυνο μη ύπαρξης διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο. Τελούμε να αναμονή σήμερα λοιπόν. Έχουμε συνεδρίωση των σκιωδών το βράδυ για το πακέτο για την ασφάλεια των προϊόντων και τον έλεγχο της αγοράς. Και περιμένουμε τι θα αποφασίσει η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων σήμερα. Ευχαριστώ. Όπως ήδη ακούσατε, δεν είναι ιδεώδης η κατάσταση. Στριμωγμένοι είμαστε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αν σκεφτούμε το περιεχόμενο του πακέτου, είναι κάτι που θα θέλαμε να περάσει. Όμως, έτσι πιστεύω τουλάχιστον, ίσως κάποια κράτη-μέλη να μην είναι τόσο πρόθυμα να προχωρήσουν με το πακέτο. Ίσως υπάρχουν εικασίες ότι μετά τις εκλογές οι ισορροπίες στο Κοινοβούλιο θα είναι διαφορετικές. και ίσως να μην υπήρχε τόσο αυστηρή πρόταση για την εποπτεία της αγοράς και ίσως αυτό να είναι σβάρος των καταναλωτών και όσον αφορά τις ισότιμες συνθήκες για τους Ευρωπαίους παραγωγούς και την εξοπλιστία της εσωτερικής αγοράς. Γι' αυτό στείλαμε επιστολή που τα λέει σταράτα και τη στείλαμε στο Συμβούλιο και θα δούμε τι θα γίνει. Είναι η θέση επαναχώρησης αυτή. Εάν δεν δούμε πρόοδο, τότε θα πάμε στην Ολομέλεια. Όμως χρειάζεται να έχουμε ένα παραθυράκι ανοιχτό. Και ίσως μπορούμε να βρούμε μέσω του ΕΛΚ κάποια μέσα πολιτικής πίεσης, να σπρώξουμε το Συμβούλιο να διαπραγματευτεί. Αυτός είναι ο απότερος στόχος, να περάσει η νομοθεσία και να ξεκινήσουμε ταχύτερο δυνατόν τις ε, διαπραγματεύσεις. Έτσι βλέπω εγώ λοιπόν την ε, όλη κατάσταση. Πρόεδρος Καλός, θα συναντηθούμε το απόγευμα, το βράδυ μάλλον, και θα κάνουμε ανακοίνωση αύριο το πρωί αναλόγως. Και αύριο να είστε όλοι εδώ για την ψηφοφορία. Εγώ ελπίζω ότι ίσως τελικά εγκριθεί η πρόταση. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξο όμως αφορά τα είδη κεραμικής βασικά, η πρόταση, που είναι φτιαγμένα στην Αγγλία βασικά. Αυτά, τα, εδώ τα κύπελα, τα φλιτζάνια, τα φτιάχνουμε στην εκλογική μου περιφέρεια, κάθε φορά πίνετε καφέ να σκεφτώσετε το stock on trend. Πρώτη ανάγνωση, της διαπραγματεύσεις στην πρώτη ανάγνωση. Έγινε άτυπη συζήτηση χθε για τη μεταφορά των οχημάτων, των οχημάτων και θα ψηφιστεί αύριο. Θέλαμε όμως προτακτικές συζητήσεις με την ελληνική προεδρία, να δούμε πώς προχωράει το πράγμα. Χρησιμότατη συζήτηση. Συζητήσαμε τα βασικά. Θέλαμε να βελτιώσουμε τη δυνατότητα των πολιτών να καταχωρούν γρήγορα και αποτελεσματικά τα οχήματά τους με ελάχιστη γραφειοκρατία. Περί αυτού πρόκειται. Τα κράτη-μέλη έχουν κολλήσει για διπλούς και τριπλούς ελέγχους των πάντων. Παρά το γεγονός ότι έχουμε έγγραφα για κοινή καταγραφή των ε, οχημάτων και στην Επιτροπή Μεταφορών προωθούμε ε, επίσης και την πιστοποίηση, ε, την αναγνώριση πιστοποιητικών οχημάτων. Θέλουμε να ξεπερδέψουμε λοιπόν με την καταχώρηση των οχημάτων. Κάποια κράτη-μέλη ανησυχούν για την καταβολή συμπληρωματικών φόρων όπως στη Δανία, έχουν το, τα υψηλότερα τέλη οχημάτων. Για να καταφέρεις το όχημά σου ε, στην Δανία προπληρώσεις και παραπάνω φόρο. Το επεξεργαζόμαστε όμως. Υπό την πεφωτισμένη ηγεσία του κυρίου Μάντελς, που δυστυχώ απουσιάζει, ίσως καταλήξουμε σε συμφωνία. Πρέπει να περιμένουμε όμως. Ωραία. Ωραία. Πάει αυτό. Πάμε σε σειρά συζητήσεων για τις διάφορες εργασίες μας και πώς προοδεύουν. Λοιπόν, κάθε συζητήση έχει περίπου ένα μισάωρο για κάθε θέμα. Έκθεση για το Solvit πρώτα απ' όλα. Ο κύριος Λέκεγκαρντ, ο είναι εδώ, έχουμε έξι συμβαστικές τροπολογίες προς συζήτηση. Οι σκιώδεις συγητές, κύριε Χάνσλικ, ο κύριος Φόξ είναι εδώ. Ποιος καλύπτει το S&D σήμερα. Η κυρία Μπέρο έρχεται. Και από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιο είναι εδώ. Α, καλημέρα. Την κυρία Γκρέμπελ. Μα ωραία, ωραία. Θα σα συστήσω αργότερα όταν μου πείτε το όνομα σα, έτσι. Λοιπόν, ο κύριο Λέκεργαρτ, λοιπόν. Τι γίνεται με του συμβιβασμού, κ. Λέκεργαρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπω είπαμε την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε, επεξεργάστηκα κάποιες συμβαστικές προτάσεις για να τακτοποιήσω κάπως το κείμενο, μεταξύ άλλων για την αύξηση ευαισθητοποίησης και το ρόλο των ενώσεων επιχειρήσεων για τη διάδοση βελτίστων πρακτικών και κάποια άλλα συναφή ζητήματα. Σωστά το είπατε Πρόεδρε. Έχουμε έξι συμβαστικές τροπολογίες. Αποφάσισα να μην γίνει συνεδρία συσκιωδών αλλά ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστέλλοντας τα σχέδια συμβαστικών προτάσεων στις σας ομάδε ομάδες προς σχολιασμό. Αυτό συμφωνήσαμε νομίζω την περασμένη φορά. Έλαβα κάποια σχόλια. Προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορούσα να πετύχω σωστή ισορροπία. Να πετύχω συμβιβαστικές προτάσεις. Εξακολουθώ να θεωρώ ότι πρόκειται περί εκθέσεως και στέλνει μήνυμα το Σύμβουλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη του Solvit. Δεν νομίζω ότι έχουμε προβλήματα μεγάλα, έχουμε ευρεία συνένεση. Αυτά είναι τα σχόλιά μου και περιμένω να ακούσω τα σχόλια των ε, συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χάνσλικ, να δούμε σκιώδης τι λένε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες μας πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση και θα προωθήσουν ακόμη περισσότερο το Solvit. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, γιατί πολλοί κόσμος ακόμα δεν ξέρει ότι υπάρχει αυτό το εργαλείο. Πολύ χαίρομαι λοιπόν που αυτό λαμβάνεται υπόψη στις συμβιβαστικές τροπολογίες. Τώρα, ας δούμε την τροπολογία που αφορά τη στενότερη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και των φορέων του Solvit. Βεβαίως και είμαι υπέρ, έχω υποβάλει προς αυτή την κατεύθυνση και εγώ μια τροπολογία. Τώρα, ποια μορφή θα έχει αυτή η συνεργασία, εδώ είμαι πολύ ευέλικτη. Η σύσταση των ομάδων εργασίας που προτείνει ο εισηγητής φαίνεται καλή ιδέα. Αν και θα έλεγα ότι αυτή η συνεργασία δεν πρέπει οπωσδήποτε να έχει αυτή τη μορφή και όχι άλλη. Καλό είναι να μην ε, είναι πολύ τυπική αυτή η συνεργασία. Τώρα για τα κέντρα Solvit, εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ των κέντρων, αλλά τα κράτη-μέλη πρέπει να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν ακόμα καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κέντρων Solvit. Τώρα, τη συμβαστική 4. Ε, την προσυπογράφω απόλυτα. Το Solvit είναι για όλους, νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό, άπαντες. Η αναφορά στις κοινωνικές ομάδες δεν περιορίζει το πεδίο εφαρμογής, αντίθετα αναδεικνύει τις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες που μπορεί να χρειάζονται το Solvit και θα φροντίσουμε ότι θα είναι διαθέσιμο το Solvit και σε αυτές. Οπότε είναι πολύ καλή ιδέα να αναφερθούν οι ομάδες αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά για την επικοδομητική συνεργασία μας μέχρι τώρα και σας στηρίζω σε όλα τα θέματα. Ευχαριστώ κυρία Ζαμπέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με βάση τις συζητήσεις και στην ΙΜΚΟ είναι σαφές ότι όλοι θέλουν να βελτιώσουν τη λειτουργία των κέντρων Solvit. Ε, έτσι θα διασφαλιστεί εμπιστοσύνη για, στην εσωτερική αγορά. Τώρα από την άποψη της εσωτερικής αγοράς επαναλαμβάνω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει αυτός ο μηχανισμός Solvit στη διάθεση των πολιτών και των επιχειρήσεων όποτε έχουν προβλήματα με τις δημόσιες αρχές ως μετακινούμενοι εργαζόμενοι ή κατά τη διάρκεια άλλων διασυνοριακών δραστηριοτήτων. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του και τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Θα ήθελα βέβαια μια μικρή αλλαγή στην πρώτη συμβιβαστική για να χωρίσω με τα θέματα επιχειρήσεων αφενός και ενημέρωσης από την άλλη. Χαίρομαι όμως που ζητούμε να υπάρχει η πρόσβαση γιατί θα πρέπει η προσβασιμότητα να προαχθεί. Γενικά ελπίζω να ε, συμφωνήσουν όλοι για την αυξημένη ενημέρωση για το Solvit. Πώς θα λειτουργήσει αν δεν είναι γνωστό μεταξύ των χρηστών. Και θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κέντρων Solvit. Βέβαια, τι θέλουμε να επιτύχουμε. Θέλουμε το Solvit να χειρίζεται τα προβλήματα που πρέπει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η συνεργασία μεταξύ των κέντρων να είναι ομαλή και οι τελικοί χρήστες να γνωρίζουν τις δυνατότητες που έχουν και να καθοδηγούνται στη σωστή κατεύθυνση. Αναφέρεται αυτό στην έκθεση όταν δηλαδή έχουν προβλήματα. Η συμβιβαστική τροπολογία για την πρόοδο του ε, Solvit και την προσπελασιμότητα είναι καλή. Θα πρέπει να πιεστούν τα κράτη-μέλη να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Να λάβουμε υπόψη μας όμως και τους υφιστάμενους μηχανισμούς ε, πριν σκεφτούμε την υποχρέωση, την, ε, το ενδεχόμενο της νομοθεσίας για να λειτουργήσει το Solvit. Τέλος, μια διευκρίνηση. Η τροπολογία 37. Πρόταση να έχουν την επιλογή τα κράτη-μέλη να έχουν περιφερειακά ή τοπικά κέντρα σόλβιτα. Από την προηγούμενη συζήτηση έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις που οδηγούν στο φόβο ότι η ύπαρξη αυτών των κέντρων μπορούν να αποδυναμώσουν τη λειτουργία του Solvit. Βεβαίως, θεμητή ανησυχία. Όμως, καταρχήν πρέπει να υπογραμμίσω ότι είναι ε, δυνητικό αν το κρίνουν σκόπιμο, θα κάνουν τέτοια κέντρα τα κράτη-μέλη σε συνδυασμό με τις άλλες δικτυακές πύλες σε, εθνικό, σε περιφερειακό επίπεδο για να είναι πιο κοντά στους χρήστες και να υπάρχει μια πιο άμεση, ένα άμεσο σημείο επαφής. Επίσης, τέτοια περιφερειακά γραφεία δεν πρέπει και δεν θα έπρεπε να κάνουν την επίλυση με την, με την τροπολογία μου πάω να διασφαλίσω ότι θα ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η επίλυση των διαφορών θα λαμβάνει χώρα σε επίπεδο δημόσιας εθνικής διοίκησης. Τα περιφερειακά κέντρα θα είναι σαν μια πύλη όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την καταγγελία ε, που μετά θα παραπέμπεται στην εθνική διοίκηση και μετά ε, ε, ε, θέματα που δεν αφορούν το Solvit θα παραπέμπονται έγκαιρα στις αρμόδιες αρχές. Ελπίζω να έχουμε λύσει την παρανόηση που προέκυψε και ελπίζω να υπερψηφίσετε και αυτή την τροπολογία. Τέλος, ο εισηγητής και οι σκιώδης έκαναν πολλή δουλειά, τους ευχαριστώ, η συνεργασία ήταν καλή και ελπίζω να μπορέσουμε τελικά να βελτιώσουμε αυτό το μηχανισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Ρούιλε, θέλετε να σχολιάστε. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τις συμβαστικές τροπολογίες των εισηγητή και επειδή ορισμένα πράγματα δεν τα έκανε δεκτά. Την περασμένη φορά είπαμε ότι θα ήταν πρόβλημα τώρα να διευρύνουμε τα καθήκοντα του Solvit αυτό δεν πέρασε, αν και υπήρχαν τροπολογίες. Σε αντίθεση με την προηγούμενη ομιλήτρια είμαι επιφυλακτική σε σχέση με τα περιφερειακά και τοπικά γραφεία Solvit. Νομίζω ότι τώρα θα ήταν αυτό υπερβολικό, θα δημιουργούσε υπερβολικό φόρτο και νομίζω ότι τα υφιστάμενα κέντρα Solvit πρέπει να γίνουν πιο γνωστά και μέσα στα, στα πλαίσια αυτών των υφισταμένων κέντρων θα πρέπει να φροντίσουμε για καλύτερη συνεργασία. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που και εγώ θα προσθέσω τις ευχαριστίες μου ε, προς τον κύριο Λόκιγκαρτ ε, και την ομάδα του. Χαίρομαι με τις συμβιβαστικέ λύσεις που προτείνει γιατί αντιμετωπίζονται έτσι τα προβλήματα της καλύτερης ευαισθητοποίησης, της ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο του Solvit. Βλέπω ότι οι τροπολογίες ε, δείχνουν ότι συμφωνούμε σε γενικές γραμμές για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την υπηρεσία αυτή. Μόνο προσοχή σε σχέση με τη συμβιβαστική 4 εγώ θέλω το Solvit να είναι προσβάσιμο από, όλα τα, από όλους τους τομείς ε, της, ε, ε, της κοινωνίας. Δεν νομίζω ότι είναι νομοθετική πρακτική καλή να το γράφουμε αυτό σε κάθε νομοθέτημα το οποίο συντάσσουμε. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε ευρεία προσβασιμότητα σε οδηγίες που έχουν να κάνουν με κάθε νομοθέτημα. Νομίζω ότι παρεκκλίνουμε από αυτό αν κάθε φορά ε, αναφερόμαστε σε ένα τμήμα της κοινωνίας ή σε κάποιο άλλο τμήμα της κοινωνίας σε κάθε νομοθέτημα το οποίο ε, δημιουργούμε. Γι' αυτό δεν διαφωνώ με το στόχο σας, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος να εξασφαλίζουμε ομοιόμορφη προσβασιμότητα ε, στις δημόσιες υπηρεσίες ο καθένας δηλαδή ε, να έχει κάτι να πει τέλος πάντων στο, στην, ε, στην ομοθεσία αυτή και στο πώς πρέπει να γίνει η, η διαδικασία. Πάντως, ε, εντάξει, μόνο σε αυτό διαφωνούμε, κατά τα υπόλοιπα συμφωνώ απολύτως με τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ο Πρόεδρος, ε, από την Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΚΤ έχουμε εδώ τον κύριο Γιόνσον που είναι τμήμα της ομάδας Πρέντεν που ε, έρχεται πολύ συχνά εδώ να μας ε, να σχολιάζει τις εκθέσεις μας. Να σας δώσω το λόγο για να μας πείτε ποια είναι η δική σας άποψη για το πώς εξελίσσεται το Solvit. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Νομίζω ότι τα περισσότερα έχουν υποθεί ήδη στις προηγούμενες συνεδριάσεις, τουλάχιστον από δικής μας πλευράς. Αναμένουμε εναγωνίως την έγκριση της έκθεσης αύριο. Και αυτά θα ήθελα να πω για την ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσω το λόγο και πάλι στον κύριο Λόκιγκαρτ για να συνοψίσει. Και θα ψηφίσουμε αύριο βεβαίως. Ναι. Αυτά θα είναι τα τελικά μου σχόλια βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους για τα σχόλια τους ε, και για την επικοδομητική εργασία ως τώρα. Απλώς μερικά σχόλια ε, σε συνέχεια όσων ακούστηκαν. Αν πάρουμε τις συμβιβαστικές τροπολογίες ε, μία προς μία, για τη συμβιβαστική ένα η ιδέα του να την χωρίσουμε σε δύο τμήματα. Δεν διαφωνώ, αλλά μέχρι τώρα δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο θέλετε να γίνει αυτό. Πώς θα μπορούσατε λοιπόν να μας... Ε, άμα θέλετε μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση γι' αυτό. Γιατί θέλω να καταλάβω για ποιο λόγο μου το ζητάτε αυτό. Δεν έχω αντίρρηση. Απλώς προτιμώ να κάνω το σωστό. Παρακαλώ λοιπόν να το σχολιάσουμε λίγο περισσότερο αυτό. Δώστε το λόγο στην κυρία Ζαμπέλα σε λίγο. Υπάρχει τίποτα άλλο που θέλετε να μας πείτε. Ναι, για την τέσσερα, στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Φόξ. Κοιτάξτε, Μήπως θα μπορούσατε να συμφωνήσετε κύριε Φόξ, αν, αν αλλάζαμε τη λέξη particular σε IE, για παράδειγμα δηλαδή. Για να μπορέσουμε να τονίσουμε αυτό που θέλουμε να πούμε. εγώ θα προτιμούσα να αναφερόμαστε σε αυτά ως παραδείγματα και να μην χρησιμοποιούμε το particularly. Ειδικά δηλαδή. Μετά το online portal, λέει ο κ. Fox, for all citizens, για όλους τους πολίτες να προσθεθεί. Για να εξασφαλίσουμε πρόσβαση ε, σε όλους τους πολίτες. Γιατί αν αρχίζετε να τα γράφετε όπως τα γράφετε τώρα, νομίζω ότι είναι ένα κακό προηγούμενο για τα νομοθετήματα. Αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε εκτός Επιτροπής, διμερώς άμα θέλετε. Εντάξει, καλή ιδέα, λέει ο κύριος Λόκεγκαρτ. Για το περιφερειακό θέμα τώρα, άκουσα την άποψη της Επιτροπής προσεκτικά. Νομίζω ότι έχουν δίκιο. Εγώ καταρχήν δεν έχω πρόβλημα να συμπεριλάβουμε κάπως ε, το θέμα της ενημέρωσης, αλλά θα ήθελα, όπως είπε και η κυρία Ρούλε και άλλοι συνάδελφοι, δεν θέλουμε να αυξηθούν τα καθήκοντα σε περιφερειακό επίπεδο. Πρέπει να είμαστε σαφέστατοι ως προς αυτό. Αλλά πέρα από αυτό, Νομίζω ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Αναμένω τη ψηφοφορία αύριο και μπορώ να συνεχίσω τη διμερή συζήτηση με τους ε, σκιώδεις μετά. Ε, κυρία Σαμπέλ, τα ίδια λέμε, Πρόεδρε, για τις περιφερειακές αρχές. Δεν λέω ότι πρέπει να τα κινηθούμε από εθνικό σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά να δώσουν τουλάχιστον τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν πληροφορίες σε περιφερειακό επίπεδο. Αν είναι εικονίδιο στο σελίδα στην οποία κλικάρουν και πάνε στο σελίδα του Solvit ή φυλάδια που διανέμονται σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, δεν ξέρω. Αυτό είναι θέμα ενημέρωσης και όχι υπηρεσία που παρέχεται σε περιφερειακό επίπεδο δεν λέω να έχουν περισσότερους ανθρώπινους πόρους σε περιφερειακό επίπεδο ή κάποιον που θα δίνει πληροφορίες. Αλλά οι περιφερειακοί φορείς θα πρέπει να έχουν κάποιο σημείο που θα δίνει πληροφορίες για το μηχανισμό Solvit. Αυτό εννοούσα όταν έλεγα περιφερειακό επίπεδο. Εγώ 17 χρόνια ήμουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και ξέρω έρχεται ο κόσμος, απευθύνεται σε εμά και είναι το επίπεδο το κοντινότερο στους πολίτες. Έχω εμπειρία τόσων ετών, ξέρω έρχεται ο κόσμος. Ανεξάρτητα από το πρόβλημά τους, ρωτάνε, ζητάνε πληροφορίες τα πάντα. Να τους δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν περισσότερες πληροφορίες στο επίπεδο αυτό που είναι κοντά σε αυτούς. Και έτσι δεν χρειάζεται να πάνε να ταξιδέψουν, να πλησιάσουν τις εθνικές αρχές και τα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους πρέπει να αναφέρουμε. Πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση. Και πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ελπίζω τώρα να τα είπα ξεκάθαρα. Συμφωνείτε με τον κύριο Φόξ, λέει ο Πρόεδρος, δηλαδή, και με τον κύριο Φόξ. Κύριε Λέκεγκαρτ, λοιπόν, ας πείτε τελευταία λέξη σαν εισηγητής. Ακούσαμε τα επιχειρήματα για μία ακόμη φορά για το θέμα το περιφερειακό μπορούμε να συμβιβαστούμε. Θα συζητήσουμε με τον κύριο Φόξ, θα δούμε αν μπορούμε να τα βρούμε. Σίγουρα έχετε ισχυρή ομάδα σκιωδών και αύριο θα έχουμε επικοδομητική ψηφοφορία και μετά θα ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μεγάλη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που την υποστηρίζουμε. Είμαστε, έχουμε τελειώσει δύο λεπτά νωρίτερα. Καλωσορίζω ένα νέο μέλος λοιπόν της Επιτροπής, νέο αναπληρωματικό μέλος, από την Πολωνία. Στη θέση του κύριου Τσασκόφσκι, ο κύριος Ρος. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην Επιτροπή. Μέλος του ΕΛΚ. Θέλετε να πείτε κάποια λόγια εν είδη εισαγωγής η σύσταση. Θέλετε να συστηθείτε, να πείτε μερικά λόγια σε όλους. Ωραία. Εν τη αυτή περιπτώση πάμε σε άλλο σημαντικότατο θέμα. Θα ψηφίσουμε από αυτού αύριο. Όχι, όχι, όχι αύριο. Αναβλήθηκε η ψηφοφόρη. Η κυρία Σαναλεβά θα πει γιατί αναβλήθη η ψηφοφορία. Έχουμε 27 συμβιβαστικές τροπολογίες προς εξέταση. Λείπουν κάποιοι σκιώδεις. Ο κ. Βαντερκάμπ εδώ είναι. Ακούει. Ο κ. Μάντερς. Μας λείπουν φιλελεύθεροι. Υπάρχει κάποιος από τους φιλελεύθερους. Δεν βλέπω κανέναν. Η κυρία Ρούλα και εγώ είμαστε εδώ. Σαν η βασική σκιώδης. Σημεία αναφοράς για κάθε θέμα. Κυρία Σενάροβα, λοιπόν, σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ε, ε, σκιώδεις και σας προσωπικά, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ ότι πρόκειται για σημαντική έκθεση και σημαντική νομοθεσία. Όσο πιο πολύ προσεγγίζουμε στο στόχο μας, τόσο περισσότερο πρέπει να σκεφτόμαστε ότι το σημαντικότερο στο e δεν πρέπει να το χάσουμε, δηλαδή ότι πρόκειται για ένα στοιχείο ασφάλειας. Σε περίπτωση τροχαίου, αυτομάτως καλεί σε βοήθεια μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Εμείς συμφωνούμε ότι θα πρέπει να συμβάλλουμε έτσι στη μείωση των θυμάτων στους δρόμους Ναι, είναι, ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες οι νεκροί από τροχέα. Υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον για πολλές πτυχές αυτής της έκθεσης. Ε, αφορά την προστασία δεδομένων, την ανοιχτή πλατφόρμα, τα ιδιωτικά ε, νούμερα κλήσης για περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο εξοπλισμός των οχημάτων. Όλα αυτά είναι σοβαρά θέματα, ιδιαίτερα σε σχέση με την προστασία δεδομένων και προσωπικών δεδομένων. Ε, θέλω λοιπόν καταρχήν να μην δίνει τη δυνατότητα το σύστημα να παρακολουθεί κανείς το ε, ακριβώς ε, κινείται το όχημα. Θα πρέπει το e-call να είναι ένα εργαλείο που αξιοποιεί τον αριθμό 112 και λειτουργεί δωρεάν για όλους τους οδηγούς στην Ευρώπη πέρα από τη μάρκα του αυτοκινήτου, ε, χωρίς να παίζει ρόλο αυτή δηλαδή. Ε, έπρεπε, όπως είπατε, να μεταθέσουμε την τελική ψηφοφορία, γιατί η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ επεξεργάζεται για το άρθρο 6 μία γνωμοδότηση που αφορά δηλαδή τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία τους ε, και τον κανονισμό 50 ε, από τη διάσκεψη των Προέδρων. Γι' αυτό έπρεπε να αλλάξουμε το, χρονικό, το χρονοδιάγραμμα για να προλάβει να συζητήσει η ΛΥΜΠΕ να ετοιμάσει τις ε, τροπολογίες ε, και κατά την τελική ψηφοφορία η Επιτροπή μας να λάβει υπόψη μας την γνωμοδότηση αυτή της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Γι' αυτό δεν θα ψηφίσουμε αύριο όπως είχε αρχικά προβλεφθεί αλλά αρχές Φεβρουαρίου. Είχα τη δυνατότητα χτες να συμμετάσχω στη συνεδρίαση των ε, σκιωδών από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και νομίζω ότι πάμε καλά. Τώρα για τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Είπαμε ήδη ότι προετοιμάσα 27 ε, συμβιβαστικές που καλύπτουν τις ε, περισσότερες από τις 123 τροπολογίες. Όμως ε, και από την Επιτροπή Τραν και Ήτρε λάβαμε ε, τροπολογίες. Ε, με τους Σκιώδης μπορέσαμε την περασμένη Τετάρτη στο Στρασβούργο να τη συζητήσουμε και χαίρομαι τις τροπολογίες τους και χαίρομαι που δεν είχαμε μεγάλα προβλήματα. Επίσης ζήτησα συμπληρωματικές γραπτές απόψεις από, τον, από τους Σκιώδης και έλαβα γνωμοδότηση μέχρι τώρα από την πολιτική ομάδα ΕΛΚ και θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Φαντερκάμπ. Τώρα, ποια είναι τα σημαντικότερα θέματα όπως υπάρχουν στις συμβιβαστικές τροπολογίες. Ένα θέμα είναι η συμβατότητα του Equal με το Γαλιλαίο και Έκνος. Αυτό υπάρχει στην τροπολογία 3 και 17. Για αυτά τα δορυφορικά προγράμματα θέλω να συμπληρώσω τη λέξη operational, λειτουργικό. Ένα άλλο είναι η συνύπαρξη ιδιωτικών συστημάτων και του δημοσίου συστήματος ECOL. Αυτή είναι η τροπολογία 16. Οι καταναλωτές θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν και ενδεχομένως να έχουν και ιδιωτικό σύστημα. Αλλά οι κατασκευαστές πρέπει να εγγυώνται ότι στο όχημα θα υπάρχει και το δημόσιο σύστημα ε, με τον ε, αριθμό 112 και θα είναι εγκατεστημένο αν δεν είναι λειτουργικό το ιδιωτικό σύστημα και θα είναι βέβαιο ότι θα ενεργοποιείται το σύστημα. Τώρα για την ανοιχτή πλατφόρμα 8, 18 και 19 τροπολογίες. Το e θα είναι ένα στοιχείο ασφάλειας και μόνο. Καλούμε όμως την Κομισιόν σε να αρχίσει διαβουλεύσεις με τους εμπλεκομένους και να συζητήσει τι απαιτήσει ε, θα πρέπει να υπάρξουν για την ανοιχτή πλατφόρμα και να υποβάλουν χωριστή ε, νομοθετική πρόταση για την πλατφόρμα αυτή και τις δυνατότητες πρόσβασης στην πλατφόρμα και τις προϋποθέσεις γι' αυτό. Τώρα, ε, ημερομηνία θέση σε ισχύ συμβαστικές 25 και 27. Θέλω να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2012 ζήτησε ε, από το 2015 να είναι υποχρεωτικό το e-call στους νέους τύπους οχημάτων από τον Οκτώβριο του 2015. Θέλουμε να τηρηθεί αυτή η προθεσμία και γνωρίζουμε ότι όλοι ε, φορείς, οι εμπλεκόμενοι ε, για την επιτυχία χρειάζονται χρόνο. Πρέπει να ε, υιοθετηθούν και οι κατεξουσιοδότηση πράξεις και γι' αυτό θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και ίσως να ξανασκεφτούμε την ε, ημερομηνία. Οι εκθέσεις αξιολόγησης, αυτή είναι η συμβιβαστική 26, εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνω να ζητήσει τρεις εκθέσεις. Η πρώτη αφορά την ε, προετοιμασία των υποδομών για να αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα και απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να μπορεί να αξιοποιείται το σύστημα. Η δεύτερη ε, έκθεση θα πρέπει να ε, γίνει το 2018 και θα εξετάζει αν ο κανονισμός μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τύπους οχημάτων. Και μετά ζητούμε έκθεση για την ανοιχτή πλατφόρμα η οποία θα πρέπει να συμβαδίζει και με νομοθετική πρόταση. Η Λίμπε στις 30 Ιανουαρίου θα ε, γνωμοδοτήσει μετά την ψηφοφορία εκεί οι Σκιώδης και όσοι, ε, θα, ε, όλοι, συμμετέχουν θα στείλουν τις τροπολογίες τους και ενδεχομένως ε, θα συγκληθεί και άλλη συνάντηση των σκιωδών. Νομίζω όμως ότι αυτή η δεύτερη συνάντηση δεν θα χρειαστεί. Μετά στην Επιτροπή ΙΜΚΟ θα γίνει ψηφοφορία για την τελική μορφή της έκθεσης και τελική ημερομηνία θα είναι η 11η Φεβρουαρίου. Αυτό προτείνω. Μετά, στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος μας, ε, που το συμφωνήσαμε μεταξύ μας και με την Τραν, θα έλεγα να πάει για ψηφοφορία στο Στρασβούργο η έκθεση στη δεύτερη ολομέλεια του Στρασβούργου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία ε, Άλοφα. Εγώ συναντήθηκα με τον πρόεδρο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, το Στρασβού, στο Στρασβούργο, και του εξήγησα ότι είμαι πολύ ικανοποιημένο με το γεγονό ότι ε, ε, μάλλον δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένο με το γεγονό ότι μόνο τόσο τελευταία στιγμή ενεπλάκησαν στη συζήτηση. Τρία χρόνια το συζητάμε αυτό και εκείνοι εμφανίζονται την τελευταία στιγμή και αν δει κανεί ε, τα θέματα τη προστασία δεδομένων θα διαπιστώσει από τι συμβιβαστικέ ε, προτάσει τη κυρία Ενάλοβα ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί να καλύψουμε και αυτά τα θέματα και του εξήγησα, εξήγησα στον πρόεδρο τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που μα υποχρεώνει δύο εβδομάδε να καθυστερήσουμε την ψηφοφορία μα για να συμπεριλάβουμε τη δική του άποψη. Δεν μπορούμε να κάνουμε όμω τίποτε, αλλά ελπίζω να μην επηρεάσει το, την πρόοδο που θα κάνουμε με το Συμβούλιο. Είναι πολύ απογοητευτικό πάντως. Να ακούσω τώρα τους κοιόδης εισηγητές για το θέμα αυτό, ο κύριος Κάμπ που ήταν πραγματικά πάρα πολύ δραστήριος για το θέμα αυτό. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ τη Γραμματεία και το προσωπικό της Επιτροπής για τη δουλειά που έκαναν και τις προσπάσεις που κατέβαλαν μέχρι τώρα. Με κάποια έκπληξη βλέπω αυτό που κάνουν οι συνάδελφοι της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Και εγώ ανήκω σε αυτή ανήκα, ανήκα σε αυτή την Επιτροπή θα έκανα περισσότερα. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ φαίνεται ότι ασχολείται πάνω απ' όλα με το θέμα του κουμπιού switch on, switch off. και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Αυτή είναι μια δυνατότητα που στην Επιτροπή μας δεν καλύπτουμε. Λοιπόν, Πρόεδρε, έχω μια ερώτηση όσον αφορά το 8, το 19 και το 27, 26 συγγνώμη. Της ανοιχτής πλατφόρμας δηλαδή το ζήτημα. Έχουμε πετύχει ένα, κάποια συμφωνία πάνω σε αυτά. Δεν μπορεί να έχει δευτερεύουσα θέση αυτή η ανοιχτή πλατφόρμα. Πρέπει όμως να κινηθεί έγκαιρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λύσει το, τα προβλήματα, τα εκκρεμή. Το 26 πρέπει να γίνει μελέτη σκοπιμότητας εκεί. Στις 8, στην τροπολογία 8 και στην τροπολογία 19 δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μελέτη σκοπιμότητας. Αυτή την έκφραση εγώ θα ήθελα να τη διαγράψουμε. Ε, διότι θέλουμε όλα να ξεκινήσουν από την αρχή. Πρέπει να το σκεφτούμε. Στο 18 αυτό αφορά ότι δεν θα είναι μόνο οι επίσημοι αντιπρόσωποι που θα επισκευάζουν τις συσκευές και τα μηχανήματα. Και έχει διαγραφεί η οχήματα, είναι σωστό αυτό. Αν διαγραφεί η λέξη οχήματα, δεν θα μπορούμε να παρεύουμε στον τομέα των αυτοκινήτων, εκτός από την επισκευή του συστήματος Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε. Οι ανεξάρτητοι επισκευαστές μέσω της διαγραφής ε, του, της λέξης οχήματος δεν θα πρέπει να τεθούν εν αμφιβόλο, να μην μπορούν να παρέμβουν. Μετά, η ανοιχτή πλατφόρμα αναφέρουμε ότι δύο χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ του κανονισμού θα εφαρμόζεται αυτό το μέτρο. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να πούμε δύο χρόνια μετά την αποδοχή του κανονισμού. Ξέρετε ότι έχουμε τον τριμερή διάλογο μετά την αποδοχή και μετά τη θέση σε ισχύ. Πρέπει να προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα. Είναι δυνατόν αυτό. Και μετά το χρονοδιάγραμμα. Ελπίζω εσείς μαζί με τη Γραμματεία να μπορείτε να εγγυηθείτε ότι θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Διαφορετικά θα έχουμε πολλά χρονικά προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτές τις παρατηρήσεις είχα. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Μάντελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις προσπάθειες που κατέβαλε. Θεωρώ ότι πρέπει να συμφωνήσουμε με τον συνάδελφο Βαντεκάμπ για το περιεχόμενο και ίσως πρέπει να αναβάλουμε κάπως την ημερομηνία ψηφοφορίας τα κατεπήγοντα, ε, ε οι κατεπήγουσες όταν λειτουργήσει το σύστημα πώς θα λαμβάνουν χώρα ε, και πώς θα κινητοποιούνται τα διάφορα μέσα διάσωσης. Και, πρέπει... Και μπορώ να σας πω ότι ειλικρινά, όσον αφορά το privacy, την ιδιωτική ζωή, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, είναι πολύ σημαντικό όταν συμβεί ένα τύχημα και ανοίγει ο αερόσακος, μπορεί να μην έχω τραυματιστεί και να κουμπίσω το κουμπί του το call ίσως να μην χρειάζεται όμως βοήθεια. Και αν δεν ανοίξει το, ο αερόσακος, ίσως μπορώ να χρησιμοποιήσω και το τηλέφωνο, το κινητό, χρειάζομαι κάποια βοήθεια. Πρέπει να δούμε λοιπόν αν η προσέγγιση είναι σωστή. Το κουμπί δεν συνδέεται τόσο με την ιδιωτική ζωή, αλλά εάν πρέπει να κληθεί ένα ασθενοφόρο, όταν πραγματικά υπάρχει ανάγκη σε περίπτωση ατυχήματο. Εκείνη που χρειάζεται να πατήσουμε το κουμπί για το e-call. Ρούλα. Ε, κυρία Ρούλε, ευχαριστώ. Θέλω να πω κάτι που δεν το αναπτύξαμε όπως πρέπει. Το σύστημα αυτό πρέπει να σώσει ζωές, να βελτιώσει την ασφάλεια. Τώρα γίνεται υποχρεωτικό. Αποφασίζει το Κοινοβούλιο υποχρεωτική εισαγωγή. Και σε κάποια κράτη-μέλη, όχι σε όλα, αλλά στη δική μου για παράδειγμα ανοίγουν νέες συζητήσεις. Αν και το Κοινοβούλιο ασχολείται δύο-τρία χρόνια πλέον με το θέμα, ε, η κοινή γνώμη τώρα ενημερώνεται. Παλιά δεν είχε ενημερωθεί ότι θα γίνει υποχρεωτικό το σύστημα. Είναι σωστό λοιπόν να προσέξουμε λίγο περισσότερο το θέμα της προστασίας δεδομένων. Και είμαι ευγνώμων στην εισηγήτρια που ανέθεσε να γίνει αυτό το briefing paper. Αυτό το ενημερωτικό έγγραφο θα δημιουργήσει το σωστό πλαίσιο, γιατί και στην ομάδα μου υπάρχουν κάποιες απορίες σχετικά με το σύστημα ε, που δεν πρέπει να περιβάλλει ε, περί τα στοιχεία. Αν θέλουμε να ληφθούν υπόψη τα θέματα προστασίας των ε, δεδομένων, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις συστάσεις αυτού του briefing paper που λέει ότι πρέπει να ορίσουμε την ελάχιστη ποσότητα δεδομένων που πρέπει να περιλαμβάνονται και θα πρέπει το ελάχιστο αυτό να οριστεί με βάση ε, την αναλογικότητα και θα πρέπει να είναι όσο πιο λίγα γίνεται τα δεδομένα. Αυτό θα πρέπει να το συνεννοηθούμε με τη ΛΥΜΠΕ για να είναι καλή συμβιβαστική λύση και θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την καλή δουλειά που έκανε μέχρι τώρα και για τον έξυπνο τρόπο ε, που αντιμετώπισε το ζήτημα της προστασίας των δεδομένων. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι οι συμβιβαστικές θα μας βοηθήσουν να ε, περάσει από την Επιτροπή η έκθεση. Όπως είπε και η κυρία Ρούιλε, αποδείξατε ότι χειριστήκατε πολύ καλά το θέμα της προστασίας των δεδομένων, πέρα από τα άλλα πολλά θέματα. και ο εισηγητής από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ πήρε πολύ ζεστά το θέμα. Το μόνο σχόλιο μου αφορά την ημερομηνία εφαρμογής. Είναι ρεαλιστικό αυτό που προτείνεται και νομίζω ότι ε, ε, αυτή είναι σύνθετη πρόταση γιατί έχουμε και τα, ε, ε τους τύπους των οχημάτων. Θα πρέπει Νομίζω πάντως ότι έχουμε μια χρήσιμη βάση για συζητήσεις Λοιπόν, θα δούμε τι θα αποφασίσει και η Επιτροπή μετά την ψηφοφορία. Ε, καλό θα ήταν να προχωρήσουμε σε μια εντολή και αν συμφωνήσουν οι σκιώδεις μπορεί να το ζητήσει αυτό στο τέλος της ψηφοφορίας αύριο. Το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε για να προχωρήσουμε με το Συμβούλιο στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Ίσως θα ήταν υπεραισιόδοξο να, έχω, να πούμε ότι θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα, αλλά θα πρέπει να έχουμε το νου μας γιατί η πρόταση είναι σημαντική και πρέπει να επιτελέσουμε πρόοδο. Είναι σημαντικό για την οδική ασφάλεια, για τους πολίτες και Όλα αυτά τώρα μας πήραν δέκα χρόνια μέχρι να τα φτιάξουμε από τότε που τέθηκε για πρώτη φορά το θέμα και υπάρχουν μνημόνια ε, συνεργασία σε διάφορες χώρες για την εισαγωγή του συστήματος. Θέλουμε λοιπόν να γίνει πρόοδος πριν ε, λήξει αυτή η θητεία του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ λοιπόν. Ο κύριος Μαρινέσκου ε, είναι μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας και είναι παρόν για να συμβάλλει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Μία παρατήρηση έχω να κάνω για τις συμβιβαστικές 3, για την αιτιολογική σκέψη 6 και τη 17 για το άρθρο 5 παράγραφος 3. Είναι η ίδια παρατήρηση όμως και για τις δύο. Αυτές οι δυο παράγραφοι ζητούν συμβατότητα με τα δορυφορικά συστήματα. Αλλά προσθέσατε στο κείμενο της Κομισιόν τη λέξη operational, λειτουργικό. Δεν νομίζω ότι είναι σωστή η προσθήκη γιατί το, ο Γκαλιλαίο δεν είναι λειτουργικό τώρα. Θα είναι στο τέλος του χρόνου ή στις αρχές του 2015. Αλλά οι προδιαγραφές για τη βιομηχανία, για τους κατασκευαστές που πρέπει να έχει συστήματα συμβατά με τον Γαλιλαίο, αυτά υπάρχουν ήδη επίσημα, είναι δωρεάν, υπάρχουν στο διαδίκτυο και η βιομηχανία μπορεί να κατασκευάσει ε, συστήματα λήψης ε, συμβατά με τον Γαλιλαίο. Αν βάλουμε τη λέξη operational, αυτό δεν είναι κίνητρο για τον κατασκευαστή να ε, κατασκευάσει συστήματα λήψη για τον Γαλιλαίο. Ενώ όλοι θέλουμε να προωθήσουμε το σύστημα Γαλιλαίο στην αγορά με τις διάφορες εφαρμογές. Και αυτό το e είναι πολύ σημαντική εφαρμογή για τον Γαλιλαίο. Ζητώ λοιπόν να διαγράψουμε τη λέξη operational. Νομίζω ότι το κείμενο της Κομισιόν είναι καλό αν θέλετε το, να διατηρηθεί το in particular δεν με νοιάζει. Αλλά να αφαιρεθεί από την παράγραφο αυτή η λέξη operational, λειτουργικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας τα λέτε όλα αυτά από τον κλάδο, γιατί παρακολουθούν και εκείνοι το Γαλιλαίο. και με το μικρό. Η κυρία Μπάρμπαρα Πανασούτο είναι εδώ νομίζω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων έχει ασχοληθεί με τα μηχανοκίνητα οχήματα για κάποιο διάστημα. Μήπως θέλετε να μας πείτε κι εσείς ε, κάποια σχόλια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Θα ήθελα επίσης ε, να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας, ε, την εισηγήτρια την κυρία Σενάλοβα και του σκιώδει εισηγητέ ε, για την σκληρή δουλειά τους, για μια πολύ σημαντική πρόταση, για την οδική ασφάλεια και του πολίτες. Όσον αφορά τις συμβαστικέ τροπολογίες, συμφωνούμε το γεγονός ότι διατηρείται η ουσία των προτάσεων ε, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, ε, όσον αφορά ε, το ότι ο κανονισμός θα έπρεπε να αφορά κυρίως τις καταστάσεις της επίγουσες μέσω που γνωστοποιούνται μέσω του 112, οι προσπάθειες που έγιναν ε, για μεγαλύτερη σαφήνεια στο κείμενο, είτε για τους ορισμούς, είτε για τις αναφορές, ε, ε, για τις ισχύουσες προδιαγραφές, μας βρίσκουν σύμφωνες. Όσον αφορά τη θέση μας για την πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης, συμφωνούμε ότι αυτή τη στιγμή θα δημιουργούσε ένα νομοθετικό κενό σε σχέση με την κυριότητα και την ευθύνη και καθυστέρη ε, στο σύστημα, στο να είναι ε, επιχειρησιακό το σύστημα ε, κλήσης του 112 και πιστεύουμε ότι θα έπρεπε οι διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς να αρχίσουν το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσουμε να ορίσουμε τις προδιαγραφές μιας ανοιχτής πλατφόρμας πρόσβασης. Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα τώρα που είναι η η εισαγωγή, στις, ε, η εισαγωγή των, ε, της συμμετοχής σε τρίτων μερών, στη, τρίτων υπηρεσιών. Μιλάω για τη συμβιβαστική τροπολογία 16. Το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες στην αγορά διαθέσιμες ε, ήδη εδώ και πολύ καιρό και έχουν φανεί πολύ χρήσιμες. Το 112 ούτως ή άλλως θα είναι υποχρεωτικό κάποια στιγμή σε όλα τα αυτοκίνητα Οπότε οι τρίτες υπηρεσίε θα είναι μια επιπρόσθετη εναλλακτική επιλογή. σω υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα έπρεπε διεξοδικά να εξεταστούν αν όντω ε, ε, συμπεριληφθούν ε, οι υπηρεσίες αυτές, ειδικότερα σε σχέση με τεχνικά ζητήματα και ειδικότερα σε σχέση με τα θέματα προστασίας δεδομένων. Σε σχέση με την προστασία δεδομένων ενδεχομένω να χρειαστεί να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο λίγο διαφορετικό από το 112 ε, δεδομένου της δεδομένης περιπλοκότητας ε, του, των συστημάτων αυτών. Και για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη διαλειτουργικότητα και ώστε ο μηχανισμός μετάβασης να είναι αποτελεσματικός και να μπορεί να εγκρίνεται ε, στην έγκριση τύπου του οχήματος. Νομίζουμε πάντως ότι υπάρχει ανάγκη να εξεταστούν κάποια τεχνικά ζητήματα και κυρίως αυτά που έχουν να κάνουν με την προστασία των καταναλωτών. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Να ε, δώσω τότε το λόγο στην κυρία Σεναλόβα, την εισηγήτρια, για να συνοψίσει και να μας πει ποια είναι η άποψή της για τα υπόλοιπα σχόλια των, σχόλια των σκιωδών εισηγητών. Ευχαριστώ πολύ όλους για τα σχόλια. Πολύ σύντομα. Να πω δύο λόγια μετά τις παρεμβάσεις σας. Κύριε Βανταρκάμπ, ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο που κάνατε. Ευχαριστώ πολύ διότι αναφέρατε αυτό το κουμπί διακοπής και τη σχετική συζήτηση. με την άποψή σας. Και εγώ νομίζω ότι εδώ πρόκειται για την ευθύνη, για τη λειτουργικότητα. Εδώ συμφωνούμε απόλυτα. Τώρα για την πλατφόρμα ανοιχτή πρόσβασης. Είμαι σύμφωνη ότι είναι πολύ περίπλοκο το θέμα, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με νομοθετική πρόταση ειδική. Αυτό σημαίνει ότι και εγώ νομίζω ότι πρέπει να επιταχύνουμε παρακαλώ την μελέτη σκοπιμότητας. Την προθεσμία, να θέσουμε προθεσμία ενός έτους. Δεν υπάρχει λόγος γιατί να είναι πιο μεγάλη προθεσμία. Τώρα, για την συμβιβαστική 18. Εδώ ε, καλύψαμε διάφορες τροπολογίες. Ίσως καλό θα ήταν να μας πει ο κυρίος Βάντερ Κάμπ αν η λέξη vehicle πρέπει να μείνει στη συμβιβαστική, αν θέλετε να παραμείνει ή να διαγραφεί. Εδώ πρόκειται κυρίως για αυτή τη λέξη στη συμβιβαστική πρόταση. Τώρα για τον κύριο Μάντερς νομίζω ότι είναι σημαντικό και το συζητήσαμε αυτό όταν συζητήσαμε για κάθε τροπολογία χωριστά. Είναι λοιπόν σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν είναι ε, σοβαρά όλα τα τροχέα ούτω ώστε να πάνε τα συνεργεία διάσωσης. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε με τη διατύπωση αν χρειάζεται ή όχι να παρέμβουν τα συνεργεία διάσωσης. Αυτό προστατεύει τα συνεργεία αυτά. Θέλουμε δηλαδή να δράσουμε προληπτικά, να μην επιβαρύνονται υπερβολικά τα συνεργεία διάσωσης ε, με ε, λάθος ε, μηνύματα. Όπως το, με τον αριθμό 112. Τώρα, κυρία Ρουίλε, ευχαριστώ για το σχόλιο που κάνατε συμφωνώ απόλυτα ε, για το, την ανάγκη ορισμού των ελάχιστων δεδομένων. Το, η λέξη ελάχιστο είναι εδώ το μέγιστο που μπορούμε να ε, προσφέρουμε, το ελάχιστο σύνολο δεδομένων. Ελάχιστο σύνολο δεδομένων που χρειάζονται τα συνεργεία διάσωσης, ούτω ώστε να είναι αποτελεσματικά στις ε, παρεμβάσεις τους. Τώρα, στον κύριο Μαρινέσκου. Μπορούμε να το ξαναδούμε το θέμα αυτό και να σκεφτούμε πάλι την πρότασή σας. Αν και είχαν υποβληθεί σχετικά με το θέμα αυτό πολλές τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Υπήρχε ένα ερώτημα του κυρίου Βαντενκάμπ συγκεκριμένα. Ε, μήπως θέλετε να πάρετε πάλι το λόγο γι' αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε κατά την άποψή μου, καλύτερα αυτό το σημείο να το δούμε κατά τη συνεδρίαση των σκιωδών. Διότι ίσως υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Τι θέλω να πω. Αν αφαιρέσουμε τα οχήματα, θα συμπεριληφθούν και οι ανεξάρτητοι επισκευαστές, όχι μόνο οι αντιπρόσωποι. Θα πρέπει να βρούμε μεταξύ μας την καλύτερη δυνατή λύση στη συνεδρίαση των σκιωδών. Καλώς, Ρε Πρόεδρος. Έχουμε μέχρι 11 Φεβρουαρίου έχουμε χρόνο να καταλήξουμε συμβαστικές τροπολογίες. Και η κυρία Σενέλοβα κάτι θα κάνει μέχρι τότε για να ολοκληρωθεί το πακέτο. Και θα δούμε και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στην Επιτροπή ε, Πολιτικών Ελευθεριών. Έχουμε προβλέψει όμως λίγο πολύ την έκβαση. Ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε στην έκθεσή μου. Οπότε θα μπω στο ρόλο του εισηγητού σας για την γνωμοδότηση. Ποιος κοιόδης μου είναι παρόν. κυρία Μπάστος, θα έρθει η κυρία Μπάστος. Ο κύριος Κρόιτσμαν είναι εδώ. Ο κύριος Έγκστρομ καταφθάνει. Κάνει τις προετοιμασίες της τελευταίας στιγμής. Και η κυρία Βανίουλ δεν είναι εδώ, αλλά και αυτή θα έρθει. 10 και 4 πρέπει να ξεκινήσουμε. Είναι 10 και 15. Άρα μπορούμε να προχωρήσουμε. Mrs. Bastos is just signing in, so we'll uh, start. Mr. Engstrom, is, his seat is vacant, and he's. Uh... Λοιπόν, μόνο η κυρία Βανιούλ λείπει για την ώρα. Όλοι οι άλλοι έχουν έρθει. Okay, well let's make a start then. Um... Ξεκινήσουμε λοιπόν. Ο Άντωνι Βίλαν και η ομάδα της DG Connect είναι εδώ. Ευχαριστούμε που παρακολουθείτε τις εργασίες μας προσεκτικότατα. Ήρθε και η κυρία Μπάστος. Θα καταθέσει η κυρία Βανίου. Βαρνιού. Ας ξεκινήσουμε. Να σας θυμίσω που βρισκόμαστε. Θα εθετήσουμε αύριο την γνωμοδότηση. Μετά θα πάει στην Επιτροπή Βιομηχανίας που θα εγκρίνει την έκθεση της 27 Φεβρουαρίου. Για προστασία καταναλωτών και σχετικές πτυχές έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα. Η ευρενή ψηφοφορία θα αποφασίσει το περιεχόμενο για την προστασία καταναλωτών που θα ενταχθεί στην τελική έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας για την ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο έχουμε ξεχωριστό κανονισμό. Η Επιτροπή Βιομηχανίας έχει μεικτή αρμοδιότητα με εμάς, κοινή αρμοδιότητα. Έχουν αρκετές τροπολογίες. Μία αφορά το 23.5, το άρθρο 23.5 που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα, παραδόξως. Αλλά θα καταφέρουμε κάπου να καταλήξουμε για τον κανονισμό για ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο. Διότι η ομάδα της Επιτροπής Βιομηχανίας ε, κινείται προς παρόμοια κατεύθυνση με μας, άρα κάπου θα καταλήξουμε. Διαδικαστικά. Τι κάναμε μέχρι τώρα. Κάναμε πολλά. Ευχαριστώ όλους τους κοιόδης για την ενεργητικότητά τους. Τους πιέσαμε αρκετά για καλούς συμβιβασμούς. Τα καταφέραμε αρκετά καλά. Βέβαια, όπως πάντα στους συμβιβασμούς δεν είναι όλοι ικανοποιημένοι. Όσον αφορά το ποσοστό περιεχομένου, η ισορροπία κλείνει προς συμβαστικές λύσεις. 90% των λύσεων που βρήκαμε είναι συνένεση. Οι σκιώδεις με έπεισαν να προσθέσω λεπτομέρειες. Υπέρ των καταναλωτών. Δεν θέλω να αναφερθώ εκτενώς αυτό. Το συζητήσαμε αρκετά σε προηγούμενες περιστάσεις. Έχουμε εκδοχή τρία των συμβιβαστικών. Έχετε τις εκδοχές ένα και δύο ήδη, αλλά έγιναν και αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Θέλω να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία που δεν συζητήσαμε για διεύρυνση της υπηρεσίας 112 και σχετικές τροπολογίες. Η κυρία Βαρνιό ε, είναι αυτή που προτείνει αυτά τα θέματα και θέλω να την ακούσω. Συζητήσουμε κάποια άλλα σημεία περιμένοντας την κυρία Βαρνιό. Διότι θέλω να της επευθύνω το λόγο για τα θέματα του 112. Ας ασχοληθούμε το μεταξύ με κάποια άλλα. Θυμηθείτε κάτι. Έχουμε συνένεση για αναδιάθρωση της πρότασης σε επίπεδο σκιωδών. Εγώ θα αναφερθώ σε τροπολογίες όσον αφορά την οδηγία καθολικές υπηρεσίες και δικαιώματα χρηστών. Άρα οι τροπολογίες αφορούν την υφιστάμενη νομοθεσία, την οδηγία. Τα κράτη-μέλη έχουν ακόμα τη δυνατότητα, βάσει οδηγίας βέβαια, να βελτιώσουν κάποιες προτάσεις αν θέλουν. Και κάποιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν αυστηρότερες διατάξεις και εμεί ε, αυτό είναι το ελάχιστο επίπεδο που ζητούμε. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν. Στις συμβαστικές συμπεριέλαβα και απόψεις των πρασίνων. Δηλαδή, για τις πληροφορίες που παρέχονται πριν τη σύναψη της σύμβασης και τις πληροφορίες που χορηγούνται τακτικά στα, στους καταναλωτές και μπορούν να προσθέσουν προτάσεις στα κράτη-μέλη και εθνική φορείς και επειδή συντονίζονται με άλλους φορείς μπορεί όλα αυτά να καταλήξουν να γίνουν βέλτιστες πρακτικές και σχετικές κατευθυντήριες. Αυτό περιλαμβάνεται σε μια συμβαστική. Για την ενημέρωση πριν την σύναψη της σύμβασης έχουμε συμφωνήσει. Συζητήσαμε τι θα γίνει αν ο τελικός ε, χρήστης δεν έχει χρησιμοποιήσει τα ταρματικά, το τελικό προϊόν, το τερματικό προϊόν, αν αγοράσουν ας πούμε ένα τηλέφωνο, μια συσκευή από άλλη χώρα, τι γίνεται. Θέλουμε ρεαλιστική προσέγγιση να φάσει υπηρεσίες παρέχονται στον καταναλωτή. Προσυμβασιακές και μετά συμβασιακές πληροφορίες. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πώς θα ενημερώνουν οι καταναλωτές. Ρεαλιστικά. Όσον αφορά την ταχύτητα σύνδεσης. Δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμα πάνω σε αυτό. Πολλές ρυθμιστικές αρχές και φορείς ε, έκαναν κάποιες προτάσεις οι ρυθμιστικοί φορείς υπερασπίζονται τη δική μου διατύπωση, δηλαδή που κανονικά διατίθεται. Normally available. Και η κυρία Βερνιό θα αναφερθεί στο θέμα. Δεν είναι ρεαλιστικό κατά την άποψή μου να πούμε επί του παρόντος διαθέσιμες. Διότι κάθε φορά πρέπει να γίνεται αξιολόγηση για κάθε καταναλωτή που ζει και τι υπηρεσίες του παρέχονται. Τι γίνεται με τον τοπικό βρόχο. συνήθως διαθέσιμα στον τόπο του τελικού χρήστη είναι μια γενικόλογη διατύπωση που βολεύει τους παρόχους υπηρεσιών. Αυτό συνοδεύεται από νέα αιτιολογική σκέψη. Το συζητήσαμε αυτό χτες. Την αιτιολογική σκέψη 56 της Οδηγίας Καθολικών Υπηρεσιών την τροποποίησα. Δίνει προσανατολισμούς περί της συνήθως διαθέσιμης ταχύτητας. Τι σημαίνει. Η Μπέρεκ θα είναι υπεύθυνη για κατευθυντήριες γραμμές και για επικαιροποίηση αυτών. Διότι αυτό που είναι συνήθως κανονικά διαθέσιμο σήμερα αλλάζει με τις νέες τεχνολογίες. Στα κινητά, στις υποδομές κλπ. Χτες, κατόπιν προτάσεων των σκιωδών, συμφωνήσαμε ότι ένα τμήμα του πακέτου για κάλυψη κινητών δικτύων κλπ. Ε, να αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη, στην αιτιολογική σκέψη. Για τη διάρκεια και τερματισμό συμβάσεων, εν γέννη συμφωνούμε. Ανέφερα την ταχύτητα μεταβίβασης δεδομένων, συναρτήσει της ενημέρωσης του καταναλωτού στα πλαίσια της οδηγίας καθολικών υπηρεσιών για έλεγχο κατανάλωσης Άλλαξα το κείμενο περαιτέρω και έτσι είναι σαφές ότι υπάρχει βασική δυνατότητα για το χρήστη να επιλέξει προκαθορισμένο ανώτατο όριο. Δεν έχει ευελιξία να θέσει το όριό του ο καταναλωτής, αλλά επιλέγει προκαθορισμένο όριο και προκαθορισμένη δαπάνη. Και όσον αφορά έγκαιρη κατανάλωση, αυτό ισχύει σε προπληρωμένη ε, υπηρεσία και υπηρεσία πληρώνεται εκ των υστέρων. Θα υπάρχουν πάντα και εκεί ε, κατευθυντήριες γραμμές. Για αλλαγή παρόχου έχουμε γενικά συμφωνία για την αλλαγή. Στα αγγλικά switching. Για το 112 χαίρομαι που ήρθε η κυρία Βαρνιό διότι ενδιαφέρεται όλος ιδιαίτερος για το θέμα και χαίρομαι που ηγείται των προσπαθειών στον τομέα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φρονεί ότι θα έπρεπε να έχει δυνατότητα να συμπεριλάβει αυτές τις πτυχές αναθεώρηση του πλαισίου. Η Επιτροπή θέλει να πιέσει όμως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει γρήγορα. Όμως, απ' την άλλη, η κυρία Βαρνιό έχει πολύ φιλόδοξους στόχους, αλλά ίσως δεν ήταν τόσο ρεαλιστική. Εγώ υπήρξα πιο επιφυλακτικός στα προτινόμενα στη συμβαστική μας τροπολογία και ελπίζω να συμφωνούν οι συνάδελφοι, να θεωρούν το αποτελεί πρόοδο. Και στη συνεργασία με τα κράτη-μέλη μπορούμε να προχωρήσουμε. Έκανα κάποιες τροπολογίες όσον αφορά το άθρο 26 προτείνει η κυρία Βαρνιού. Και λαμβάνοντα υπόψη τα σχόλια του κυρίου Κρόιτσμαν. Και για τους δείκτε επιδόσεων, ξητικές συστάσεις, ανέφερα κάτι. Πρέπει να εμπλακούν και αρμόδιες αρχές. Αυτό δεν μειώνει όμως την εξουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και έκανα κάποια πρόταση τελευταία στιγμής μου άρεσε το σύστημα αντιστρόφου 112. Δεν ήθελα όμως να τεθεί προθεσμία να εφαρμοστεί όπως ήθελε η Μπερναντέτ, χωρίς να υπάρχει σχετική ανάλυση και αξιολόγηση συνεπιών. Πρότεινα συμβιβαστική, ζητώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε μελέτη σκοπιμότητας για το σύστημα επικοινωνιών αντιστρόφου 112 και να κάνει σχετικέ προτάσεις. Ο κύριος Βίλαν και οι συνάδελφοί του ίσως μπορούν να το αναλύσουν. Λοιπόν, θέλουμε αυτό το σύστημα σε κοινοβούλιο να το προωθήσουμε. Το αντιστρόφω 112. Αν δέχεται η κυρία Βαρνιό μια κάποια μείωση των φιλοδοξιών, θα μπορούμε να προχωρήσουμε, γιατί θα εκφράζεται έτσι η πλειοψηφία των μελών. Εξετάστηκαν πολλές λεπτομέρειες συμβιβαστικές. Γι' αυτό είμαι εκτενή στην παρουσίασή μου. Συζητήσαμε εκτενώς τις αναθεωρήσεις των διατάξεων για την ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο. Βασικός στόχος εδώ, βασικοί στόχοι, συμπεφωνημένοι, υπάρχουν. Περιπλοκότατα νομικά ζητήματα ανακύπτουν και ο καθένας έχει την άποψή του. Με τα χαράς παρουσιάζω τις σχετικές συμβιβαστικέ μου. Πέτυχα πιστεύω καλή ισορροπία. Θα διαφέρει η άποψη της Επιτροπής Βιομηχανίας, άρα θα συνεχιστούν οι συζητήσεις. Προοδεύουμε όμως για την στήριξη από πλευράς πλειοψηφίας. Στήριξη των συμβιβαστικών. Και έτσι θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσει με την Επιτροπή Βιομηχανίας, κάτι που θέλω. Έκανα προτάσεις για αλλαγέ για το άρθρο 23.5, που αφορά αποκλειστική τους αρμοδιότητα. Θεωρώ όμως ότι δεν μπορούμε να ετοιμάσουμε πακέτο χωρίς να λάβουμε υπόψη το άρθρο 23.5 και η Επιτροπή Βιομηχανίας σίγουρα με τα χαρά θα συνεργαστεί από αυτού. Η κυρία Πιλάρ Καστίγιο και μαζί μας, θα συμπεριλάβουμε δικές συμβαστικές και θα εμπλακώ στις συζητήσεις προφανώς με την Επιτροπή Βιομηχανίας. Και οι μου πιστεύω με τα χαρά σας συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις. Αυτή ήταν μια σύνοψη της καταστάσεως, κάλυψα τα βασικά, με τα χαράς να ακούσω τη δράση σας. Όσον αφορά την αυριανή ψηφοφορία, θα είναι περίπλοκος ο κατάλογος. Είχαμε πολλές τροπολογίες. Αυτό δείχνει ενδιαφέρον βέβαια. 300 τροπολογίες είχαμε τους Κιώδης και από άλλα μέλη έκανα ότι μπορώ να λάβω υπόψη περισσότερες. Αρκετές από αυτές συνεπώς θα καταπέσουν, για κάποιες συμφώνησα ξεχωριστές ψηφοφορίες για συμβαστικές. Δεν μου ικανοποιείται ότι με αυτό, όμως επειδή έχουμε πολύ μακροσκελείς περίπλοκες συμβαστικές, έπρεπε να κάνω υποχώρηση και την έκανα. Άρα κάποιες ψηφοφορίες θα αφορούν συμπληρώσεις ή κατά τμήματα ψηφοφορίες συμβιβαστικές. Διότι εν γέννη συμβαστικές έχουν γίνει αποδεκτές. Σε άλλους τομείς, αρκετούς τομείς, συνέστησα απόρριψη των περισσότερων προτάσεων που δεν αφορούν άμεσα τον τομέα ευθυνών. Η Επιτροπή Βιομηχανίας ασχολείται με αυτά. Με την περιαγωγή, παραδείγματος χάρη, Κάποιοι έκαναν συστάσεις που ακολουθούν αυτά που θέλει η κυρία Ντεκαστήγιο, κάτι που υποστηρίζω. Πολιτικός πώς συστήνω υποστήριξη της κυρίας Ντεκαστήγιο, της γραμμής της. Άρα εκεί στις τροπολογίες σας βάζω συν. Για κάποιες άλλες τροπολογίες θλίψους λέγω ότι δεν μπορώ να τι υποστηρίξω. Διότι δεν ανήκουν στη βασική μας αποστολή. Προφανώς αύριο θα ψηφίσουμε. Και αν η ομάδα, τα μέλη της ομάδας πείσουν άλλους, κάποιες θα περάσουν. Αυτό είναι το σχέδιο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση με τους Σκιώδης. Η κυρία Μπάστος ξεκινάει. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ εισηγητά για την έξοχη δουλειά που έγινε, ήταν υπέροχη δουλειά. Όσον αφορά το θέμα αυτό, έξοχη συνεργασία μεταξύ όλων των σκιωδών επαναλαμβάνω τη σημασία του ρόλου που έπαιξε ο καθένας, κάθε σκιώδης συγγητής στην προσπάθεια και θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες για τις προσπάθειες τους. Ακούσαμε μία λεπτομερέστατη παρουσίαση από πλευράς Προέδρου και εγώ θα είμαι συνοπτική. Είμαστε στην τελική ευθεία. Και Σημαντική είναι η άποψη του συγητού. 18 συμβαστικές έχω προτείνει για βασικά θέματα. Τα δικαιώματα των καταναλωτών και την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο. Αυτή η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ευαίσθητη, το ξέραμε την αρχή, όσον αφορά τον χρονισμό που θέλουμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας σαν Επιτροπή, εγκαίρως. Το χρονοδιάγραμμά μας δεν υπονομεύει την ποιότητα των εργασιών και των λύσεων τεχνικής φύσεως και νομικής φύσεως που εμπεριέχονται στη γνωμοδότηση. Πρόκειται περί θέματος μεγίστου τεχνικού εύρους. Απαιτεί λοιπόν ε, προσοχή όσον αφορά τη θέσπιση νομοθεσίας ανταποκριθήκαμε στο ύψο των περιστάσεων και μα κατήφθηνε προ σωστή κατεύθυνση ο εισηγητή. Σαν σκιώδη μπορέσαμε να παρουσιάσουμε τροπολογίες και σίγουρα ε, θα δούμε την έκβαση στην τελική ψηφοφορία. Ε, εν γέννη το κείμενο θα υποστηριχθεί, ευρέως πιστεύω. Παρουσιάστηκαν λοιπόν τροπολογίες ε, προτάθηκαν κάποιες τροπολογίες που δεν έγιναν αποδεκτές. Υπήρξαν τροπολογίες που δεν αφορούσαν απόλυτα σχετικά ζητήματα και δεν συμπεριελήφθησαν ίσως στο κείμενο, στις συμβαστικές τροπολογίες. Κάπου θα γίνουν και ξεχωριστές ψηφοφορίες για να διευκρινιστούν κάποια σημεία Στη γνωμοδότηση ενισχύονται τα δικαιώματα των Ευρωπαίων καταναλωτών, η ενημέρωσή τους λαμβάνεται υπόψη, είναι πιο αυστηρή η ενημέρωση, είναι αυστηρή, πιο αυστηρή νομοθεσία για την ενημέρωση των καταναλωτών, βελτιώνεται η διευκρίνηση α, των πληροφοριών, παίζει μεγαλύτερο ρόλο η Μπέρεκ όσον αφορά την ενημέρωση των καταναλωτών, ε, δίνουμε τη δυνατότητα στον καταναλωτή να μπορεί να ελέγχει δωρεάν την κατανάλωσή του και στις προπληρωμένες συμβάσεις και στις άλλες συμβάσεις που πληρώνονται εκ των υστέρων οι ομαδοποιημένες προσφορές ή τα πακέτα λαμβάνονται υπόψη και ίσως σε κάποια πακέτα κάποιο προϊόν να μην είναι τόσο ποιοτικό και να θέλει κανείς να διακόψει τη σύμβαση Λοιπόν, θέλουμε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η μεταφορά του αριθμού τηλεφώνου θέλουμε να καλύπτεται και το χρονικό όριο εντός του οποίου μπορεί να γίνει η μεταφορά και να υπάρχει εγγύηση δυνατότητα μεταφοράς. Όλα αυτά είναι στοιχεία πολύ σημαντικά προ συμφέρον του καταναλωτή. Αυτή η δυνατότητα μεταφοράς θα πρέπει να μπορεί να γίνεται εντό 24 ωρών και ο νέος πάροχος των υπηρεσιών θα είναι υπεύθυνος για την μεταφορά του αριθμού τηλεφώνου στο νέο πάροχο θα εγγυάται την πλήρη ενημέρωση πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταφοράς. Ε, σαφείς οι πληροφορίες για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο και στην, στις εξειδικευμένες επίσης υπηρεσίες που παρέχονται όσον αφορά το διαδίκτυο. Μετά έχουμε κάποιες στοιχείες όπως είναι ο όγκος, η ταχύτητα των δεδομένων, ε, συμπληρωματικές υπηρεσίες, το θέμα της ουδετερότητας του διαδικτύου επίσης, του δικτύου, συμπληρώθηκε στο κείμενο αυτό, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία σύγχυση, να μην πέσει θύμα ο καταναλωτής κάποιας διάκρισης. Διευκρινίζονται λοιπόν διάφορα σημεία. Να μην είναι θύμα περιορισμών ούτε παρέμβαση όσον αφορά το περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Και απ' την άλλη, οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι ευρείες και κάποιοι ενδεχόμενοι περιορισμοί θα πρέπει να καλύπτονται συμβασιακά. Η κίνηση θα πρέπει να επιτρέπεται με έναν τρόπο ώστε να μην δημιουργείται συμφόρηση στο διαδίκτυο όσον αφορά την κυκλοφορία, ίσως αν παραστεί ανάγκη και με παρέμβαση νομική. Όσον αφορά τους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς, όλα πρέπει να διευκρινίζονται. Οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς υπέχουν υποχρέωση ελέγχου της σωστής διαχείρισης της κυκλοφορίας στο διαδίκτυο. Είχαμε κάποιες, αμήμπο διαφωνία, όσον αφορά ποια λέξη θα χρησιμοποιείτε στο κείμενο για να υπάρχει αυτή η εγγύηση της κυκλοφορίας όμως η διατύπωση που χρησιμοποιείται τελικά είναι καλή να μην υπάρχει να μην δημιουργείται πρόβλημα όσον αφορά την κυκλοφορία από πλευράς εθνικών ε, παρόχων και εθνικών φορέων. Περιμένουμε ακόμα κάποιες βελτιώσεις, κάποια ρύθμιση λεπτομεριών που προανήγγειλε ο εισηγητής μας ο κ. Χάρμπουρ. Είμαι σίγουρη όμως σαν ΕΛΚ ότι το αποτέλεσμα των εργασιών είναι καλό και ότι μπορούμε να συνοδέψουμε το περιεχόμενο της τελικής γνωμοδοτήσεως που θα ψηφίσουμε αύριο μέχρι το τέλος της διαδικασίας χωρίς άλλους δισταγμούς. Ευχαριστώ. Well, thank you very much Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας και για την υποστήριξή σας. Μπερναντέτ Βερνιό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική η δουλειά του και είμαι ικανοποιημένη, όπως είπε και η κυρία Πάστος, με την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε κατά την επεξεργασία αυτής της, αυτού του συμβιβασμού όλοι επέμειναν ε, στην ε, δομή ε, της οικουμενικής οδηγίας όπως είχε προτείνει ο κύριος Χάρμπουρ, μια πιο συνεκτική δηλαδή προσέγγιση γιατί νομίζω ότι πραγματικά έγιναν σοβαρές, έγινε, σοβαρές, έγινε σοβαρή, σοβαρή πρόοδος Είχα πει μάλιστα ε, να συμπεριλάβει όλη αυτή την εξέλιξη που ούτως ή άλλως είχε γίνει στο πλαίσιο της πρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να την προχωρήσει ακόμη περαιτέρω. Νομίζω ότι λάβαμε υπόψη επίσης ε, την ε, ταχύτητα της σύνδεσης, ε, την προστασία κατά των καταχρηστικών συμβάσεων, πρόσβαση σε υπηρεσίες γενικότερης πρόσβασης και δωρεάν, μη διάκριση, κάτι το οποίο μας βρίσκει σύμφωνους και άλλωστε συμφωνεί και η Επιτροπή Ήτρε με αυτό και επίσης ε, σαφής ορισμός της πρόσβασης στο ίντερνετ και των εξειδικευμένων υπηρεσιών. Δύο σημεία μόνο δεν μας έχουν βρει ε, σύμφωνους και θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε αυτά. Πρώτον, η δυνατότητα ε, διακοπής μια σύμβαση μετά από έξι μήνες νομίζω ότι όχι μόνο μπορεί αυτό να βελτιώσει τον ανταγωνισμό αλλά πρέπει και να ξεπεράσουμε την ε, τρέχουσα κατάσταση, δηλαδή 24 μήνες ε, κατά μέγιστο και 12 μήνες ε, κατελάχιστον. Μήπως μία προειδοποίηση ενός μηνός σε περίπτωση διακοπής σύμβασης εντός 6 μηνών είναι παρκές, ρωτάω τον κύριο Χάρμπουρ να μου απαντήσει. Μάλκολμ, δίκιο έχεις όταν λες, γιατί εδώ και πολλά χρόνια που είμαι εδώ Ξέρετε ότι το 112 το υποστήριξα πάρα πολύ όσον αφορά τον εντοπισμό των, ε, κλεισο, των κλήσεων επίγουσας ανάγκης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι ασήμαντο, πρέπει να εξασφαλίσουμε την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον ορισμό των κριτηρίων εντοπισμού. Γιατί τι συμβαίνει η αρμοδιότητα, ε, της, η ευθύνη της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν είναι σαφώς καθορισμένη. Πετάνε τον μπαλάκι από τα, κράτη-μέλη στην Κομισιόν και η Κομισιόν στα κράτη-μέλη και δεν μου φαίνεται ότι αυτό είναι σωστό. Αν θέλει η, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνέχεια να υποβάλει ένα άλλο κείμενο, δεν βρίσκω ότι αυτό είναι ασύμβατο με το κείμενο που συζητούμε τώρα έχουμε καταφέρει να βρούμε τις τεχνικές βάσεις για το e-call. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα τώρα πολιτικής βούλησης πλέον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα και να ζητήσουμε καθαρά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει στον τομέα αυτόν. Δεν ξέρω αν θα μου απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω μέχρι αύριο να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε μάλλον με αυτά τα δύο σημεία. Κατά τα άλλα, είμαι απολύτω ικανοποιημένη με τη δουλειά που κάναμε υπό την ηγεσία του Προέδρου και εισηγητή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. με τις συμβιβαστικές για την ουδετερότητα δικτύων έχουμε καλή βάση και για την Επιτροπή Ήτρα και για όλο το Κοινοβούλιο. στην σημερινή αγορά είναι σημαντικό να λαμβάνει αποφάσεις ο καταναλωτής ε, εφόσον θα είναι ενημερωμένος. Ε, γι' αυτό φροντίζουμε στις συμβιβαστικές, να είμαστε όμως και ρεαλιστές. Ε, αυτό το καταφέραμε. Βοηθούμε ε, να υπάρχει σε ε, ικανοποιητική ταχύτητα πρόσβαση στο διαδίκτυο. Είναι ε, βέβαια αυτό δύσκολο να επιτυγχάνεται πάντοτε λόγω πολλών μεταβλητών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι καλό που στηρίζομαι αυτές τις τροπολογίες ε, σχετικά με την ενημέρωση και τις κατευθυντήριες γραμμές που θα ε, επεξεργαστούμε για τον ΠΕΡΕΚ. Ε, γενικά είναι ικανοποιητικό οι τροπολογίες, αν και δεν ικανοποιούνται 100% όλοι. Νομίζω ότι θα έχουμε την υποστήριξη των πολιτικών ομάδων. Για μένα είναι ουσιώδες ε, από τη μια να διαφυλάξουμε την ουδετερότητα των δικτύων, να μην υπάρχουν διακρίσεις. Ε, από την άλλη πλευρά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα όσοι παρέχουν τηλεπικοινωνίες να αναπτύσσουν ε, καινούριου τομείς ε, διότι κάνουν μαζικές επενδύσεις ε, στις τηλεπικοινωνίες. Θα γίνει αυτό τα επόμενα χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Γερμανία η υπόσχεση ήταν ε, να επενδύσει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ένα δις στα δίκτυα, ταχαία δίκτυα και τώρα δεν υπάρχουν τα χρήματα. Αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες ε, στην ε, Γερμανία και στην Ευρώπη γενικότερα πρέπει να κάνουμε, να, να ε, εξασφαλίσουμε επενδύσεις από εκείνους που δραστηριοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες και θα πρέπει ε, όλοι να κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις. Να, εμείς έχουμε κάνει καλή προπαρασκευαστική εργασία και σε συνεργασία με την Επιτροπή Βιομηχανίας. Ευχαριστώ τους ε, Σκιώδης και τον Μάλκολμ Χάρμπορ τον εισηγήτη. Τέλος, να ευχαριστήσω θερμά τους συνεργάτες της γραμματείας της ΙΜΚΟ που δούλεψαν κάτω από μεγάλες χρονικές πιέσεις. Ε, χωρίς εκείνους δεν θα τα είχαμε καταφέρει τόσο γρήγορα να ασχοληθούμε με αυτή τη σύνθετη ε, πρόταση και να καταλήξουμε και σε εξαιρετικές λύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κρίστιαν ε, Έγκστρομ. Ευχαριστώ καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ όλους. Ο εισηγητής έκανε πολύ καλή δουλειά. Η συζήτηση αυτή έγινε επικοδομητική. Είχαμε τεράστιες χρονικές πιέσεις ε, λόγω της απόφασης της Κομισιόν να παρουσιάσει αυτό το τεράστιο πακέτο στο τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας, ε, αλλά παρόλα αυτά η δουλειά έγινε πολύ καλά. Τώρα, προστασία καταναλωτών. Μιλάμε για προσυμβατικές ε, πληροφορίες, ε, έλεγχος κατανάλωσης, αλλαγή κλπ. Έχουμε καλό πακέτο εδώ. Δεν ξέρω αν ε, ομόφωνα συμφωνούμε ή αν είναι πολύ μεγάλη πλειοψηφία, πάντως εμένα με καλύπτει αυτό το κομμάτι. Τώρα για την περιαγωγή. Συμφωνώ με την κυρία Τούν ότι οι χρεώσεις περιαγωγή ιδιαίτερα στα κινητά, είναι πολύ ψηλές και αυτό βλάπτει την εσωτερική αγορά. Δεν μπορούμε να μιλάμε για εσωτερική αγορά αν δεν μπορούν οι επιχειρηματίες να χρησιμοποιήσουν στο smartphone ε, το διαδίκτυο διασυνοριακά. Ε, συμφωνώ με την κυρία Τούν ότι πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό. Δεν ξέρω αν έχουμε την πλειοψηφία για κάτι ριζοσπαστικό σε ό,τι αφορά τις χρεώσεις του, της περιαγωγής όσο γίνεται πιο γρήγορα ας κάνουμε, θα κάνω μια τελευταία προσπάθεια απευθύνω έκκληση σε όλους τους συναδέλφους να το ξανασκεφτούν το θέμα γιατί έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι για το, η περιαγωγή πρέπει να το κάνουμε θα δούμε τώρα η ουδετερότητα των δικτύων, αυτό είναι το μεγάλο θέμα, πολύ σημαντικό πραγματικά. Το διαδίκτυο είναι το πιο καταπληκτικό πράγμα μετά την τυπογραφία στην ιστορία. Ε, οι επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργούν στην Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο. Είναι κέρια σημασία ε, η αρχή της ουδετερότητας των δικτύων να διατηρηθεί η δικτυακή ουδετερότητα. Ε, να υπάρχουν ειδικέ. Ε, να, να μην ε, δώσουμε την... να, μην υπάρχει δυνατότητα να εισπράττουν χρεώσεις για διαφορετικές υπηρεσίες. Είναι πολύ μεγάλη ευρεία η πλειοψηφία από ό,τι φαίνεται στην Επιτροπή μας ε, υπέρ αυτής της ε, προσέγγισης. Τώρα Έχουμε μεγάλη υποστήριξη για την αρχή, για το θέμα αρχής τώρα. Πρέπει να φροντίσουμε και οι ορισμοί και οι διατυπώσεις στα άρθρα να είναι απόλυτα σαφείς ούτω ώστε οι έξυπνοι δικηγόροι να μην μπορούν να βρουν παραθυράκια για να υποσκάψουν τη δικτυακή ουδετερότητα μέσα από ειδικέ υπηρεσίες. Αυτό είναι το, η μεγάλη μου ανησυχία. Γνωρίζω ότι οι δικηγόροι είναι πολύ έξυπνοι άνθρωποι και αυτό είναι καλό για εκείνους, αλλά για μας σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί. Θα κάνουμε και άλλη συζήτηση σήμερα εδώ πάνω σε αυτά. Πάντως ε, πάμε να τελειώσουμε για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες. Φαίνεται να υπάρχει συμφωνία Δεν θα πρέπει δηλαδή να είναι υποκατάστατο του διαδικτύου αυτό και θα πρέπει να είναι ένα χωριστό σύστημα που θα έχει ε, αυστηρό έλεγχο. Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που όλοι, μάλλον τα ε, τα παραδείγματα που έχουν νόημα είναι ότι αν κάποιος ε, θέλει ε, με το διαδίκτυο να έχει συνδεδεμένη και τηλεόραση ή αν μια μεγάλη επιχείρηση θέλει ένα δίκτυο ενδοεπιχειρησιακό. Εδώ δεν έχουμε πρόβλημα. Στο βαθμό που αυτό δεν βλάπτει, δεν παραβλάπτει τη διαθεσιμότητα του κανονικού διαδικτύου και στη συμβιβαστική τροπολογία 11 μαζί με τη συμβιβαστική 13 Όπως είπα δεν θα δεσμευτώ οριστικά αλλά έχω την εντύπωση ότι όλοι το ίδιο θέλουμε και θα πρέπει απλώς να φροντίσουμε για την ε, πολύ προσεκτική διατύπωση. Άρα λοιπόν μάλλον ε, με κάποια νότα αισιοδοξία ε, τελειώνω την παρέμβασή μου. Ο εισηγητής έκανε εξαιρετική δουλειά και ελπίζω και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε ε, το θέμα αυτό και να συγκεντρώσουμε μεγάλη πλειοψηφία υπέρ του πακέτου. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σα Ε, περιείχονται πολλές λεπτομέρειες αυτά που είπατε. Η Επιτροπή βιομηχανία και εμεί έχουμε και άλλο κύριο συζητήσεων μπροστά μα. Άλλους δύο αγορητές έχω, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει. Κύριε Βανχάικο πρώτα, κύριε Γκαλό, κυρία Τούν και κυρία Στάιντερ. Έχουμε χρόνο, αλλά ας είστε σύντομοι, γιατί θέλω να ακούσω κι άλλους. Κυρία Βανχέλ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Μάλκομ. Ευχαριστώ για τις καλές συμβιβαστικέ τροπολογίες μετά την τελευταία μας συζήτηση. Νομίζω ότι με την αιτιολογική σκέψη διευκρινίζονται τα πράγματα. Ε, για τα κινητά δεν είχαμε πρόβλημα, αλλά για τη σταθερή σύνδεση και εκεί θα πρέπει να ε, διευκρινίσουμε τι, ε, ποια είναι η διαθεσιμότητα. Με ενδιαφέρει και η προστασία του καταναλωτή που ε, ορίζεται ποια είναι, ποιες είναι οι συνήθεις περιπτώσεις. Πρέπει και εδώ να υπάρχει διαφάνεια, ούτως ώστε ο πελάτης να παίρνει αυτό που έχει ζητήσει και όχι μια μικρότερη υπηρεσία. Ε, τώρα διευκρινίζεται όπως σας είπα η αιτιολογική σκέψη. Νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν να διευκρινιστεί το θέμα και στο άρθρο. Αλλά αν γίνεται η διευκρίνηση μέσω της αιτιολογικής σκέψης, συμφωνώ με τη συμβιβαστική τροπολογία. Εκεί που δεν καλύπτομαι είναι στην τροπολογία 11 ορισμό εξειδικευμένων υπηρεσιών, γιατί σε αυτό το σημείο Συμφωνώ με τον κύριο Έγκστρομ. Πρέπει να είμαστε πολύ ε, ακριβείς για να μην υπάρξουν παραθυράκια και να μην γίνει κάτι που δεν ε, ε, θέλαμε. Κάτι αθέμητο. Καλό θα ήταν λοιπόν να υπάρξει μια τροποποίηση, νομίζω έχει ενημερωθεί η γραμματεία, να μπει ένα εδάφιο στη, ακόμη στη συμβαστική τροπολογία πίσω από το να, να, να διασφαλίσουμε το κατάλληλο επίπεδο ποιότητας ε, του δικτύου ε, με βάση τον έλεγχο και τώρα προσθέτω για να διασφαλίσουμε ε, ε, βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα ελέγχονται από άκρου Ε, θα έχουμε το κλειστό δίκτυο Εκεί υπήρχαν κάποιες παρανοήσεις σχετικά με το τι εννοείται, αλλά με αυτό τον ορισμό, την προσθήκη, θα ε, ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες. Θα ήθελα όλες οι πολιτικές ομάδες να, μας να υποστηρίξουν αυτή την ε, προσθήκη για να μην έχουμε παράθυράκια. Νομίζω ότι γραπτός έχει υποβληθεί και στη γραμματεία. Καλό θα ήταν να ε, μπει κάπου στη συμβιβαστική. Ευχαριστώ για την συνεργασία έχουμε καλή βάση για να συζητήσουμε και με την Ήτρο ε, για τα περαιτέρω. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι αργά τώρα να βάλω οτιδήποτε μέσα στι συμβιβαστικέ τροπολογίε, αλλά πάση περιπτώσει. Άμα τα καταφέρουμε, θα μπούμε και σε διαπραγματεύσει με την Επιτροπή βιομηχανία. Και η κυρία Τελκαστήγη ούτως ή άλλως ε, επεξεργάζεται συμβιβαστικές τροπολογίες. Ελπίζω ότι στο τέλος ε, θα έχουμε μια καλή συμβιβαστική λύση. Κανείς δεν έχει το μονοπόλιο της σοφίας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ παρεμβαίνω ως, ε, συντάκτη, ως συντάκτρια γνωμοδότηση στην Επιτροπή Νομικών. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά που κάνατε με τους κοιόδης συζητητές στο πλαίσιο αυτής της ε, Επιτροπής. Θα ήθελα ενημερωτικά να σας πω ότι η έκθεσή μου, η γνωμοδότησή μου εγκρίθηκε χθες, 21 ε, Ιανουαρίου, στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και εξακολουθώ να είμαι δυσαρεστημένη με το χρονοδιάγραμμα που μας επιβλήθηκε για την ε, έγκριση της συγκεκριμένης ε, έκθεσης ε, με πολύ μεγάλη βιασύνη. Δεν είναι συνθήκε αυτέ να δουλεύουμε. Ο συνάδελφος Έγκστρομ ήταν εχθές ε, στην ψηφοφορία. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη ψηφοφορία σε σχέση με τα ιδιωτικά, τα αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης ήταν τόσο σημαντικό που στο τέλος ε, πέρασε μόνο με μία ψήφο ε, η δική μου έκθεση, παρά το γεγονός ότι οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι δεν ήταν εχθρικοί, απλώς ήταν τόσο μεγάλη ένταση για το προηγούμενο θέμα, κανείς δεν είχε μυαλό να ψηφίσει μετά. Τέλος πάντων, ε, επικεντρώθηκα σε τρία σημεία και σας το λέω απλώς ενημερωτικός. Πρώτο θέμα για την ε, άδεια χρήσης ε, μόνο ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ προτείνω ένα μοντέλο εναρμονισμένης κοινοποίησης, κατάργηση του κεφαλαίου 2 και την τροποποίηση της οδηγίας του 2002 για την αδειοδότηση. Δεύτερο, ουδετερότητα του διαδικτύου. Το έχουμε συζητήσει βεβαίως. Είπα ότι ήμουν υπέρ ε, της εισαγωγής εξειδικευμένων υπηρεσιών υπό τον όρο ότι η ποιότητα, του, η ποιότητα δεν θα ε, επηρεαστεί. Τρίτον, που λιγάκι διαφωνώ μαζί σας, είναι τα δικαιώματα των τελικών χρηστών. Πρότεινα τη διαγραφή των άρθρων 25 έως 30, γιατί η πλήρης εναρμόνιση δεν είναι ευνοϊκή για όλους τους καταναλωτές και έχω υπόψη μου για παράδειγμα τους Γάλλους καταναλωτές που θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να ε, έχουν καλύτερη απόδοση αν γίνεται Επαναλαμβάνω λοιπόν ε, αλλαγή της τροπολογίας 2002 για τις οικουμενικές υπηρεσίες και την ενημέρωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Αυτά είναι τα ενημερωτικά στοιχεία που θα ήθελα να σας υποβάλω. Ευχαριστώ πολύ. Μα νομίζω ότι συμφωνούμε τελικά. Δεν είναι πλήρω εναρμονισμένη η οδηγία, οπότε νομίζω ότι συμφωνούμε και μάλιστα απολύτως και ως προς το τρίτο θέμα. Αλλά περιμένουμε κι εμείς ε, την ε, δική σας διατύπωση όσον αφορά την ανοιχτή πρόσβαση στο ίντερνετ. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο μέχρι την αυριανή ψηφοφορία, αλλά πάση περιπτώσει θα το συμπεριλάβουμε στον κατάλογο των ψηφοφοριών μας. Α, όχι. Α, μάλιστα. Ούτως ή άλλως όμως θα λάβουμε υπόψη την γνωμοδότησή σας. Ε, Κυρία Τούν. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θα ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους ε, που συνεχάρισαν τον εισηγητή τον Μάικλ Χάμπερ. Βλέπουμε το βαθμό της καλής και επικοδομητικής συνεργασίας γύρω από το έγγραφο αυτό, που πραγματικά προκαλεί πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση. Μου φαίνεται πάρα πολύ καλό το συμβιβαστικό κείμενο. Έχω όμω κάποιες επιφυλάξεις, ειδικότερα όσον αφορά τις εξειδικευμένε υπηρεσίε. Τροπολογία 11. Έχω την εντύπωση ότι ο ορισμός του άρθρου 2 θα πρέπει να είναι λίγο πιο συγκεκριμένος. Θα έπρεπε να είναι μάλιστα κλειστός ορισμός. Δεν μπορούμε να λέμε ότι τα πάντα μπορούν να αποτελούν εξειδικευμένη υπηρεσία. Για μένα θα πρέπει να υπάρχει ένας ορισμός που να δείχνει σαφέστατα ότι μια εξειδικευμένη υπηρεσία είναι μια υπηρεσία που βασίζεται σε παραδοσιακή υπηρεσία διαδικτύου και δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθεί. Επίσης πρέπει να μιλάμε και για κλειστά δίκτυα και επιμένω μπορεί να υπάρχουν και άλλες ε, διατυπώσεις, αλλά πρέπει να αναφέρεται ότι είναι μια υπηρεσία διαφορετική από την ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο. Είναι πάρα πολύ καλή πρόταση βέβαια. Έχω υποβάλει τροπολογίες που προτείνουν να μην υπάρχουν για την περιαγωγή επιπλέον τέλη και, η την εναρμόνιση από τον Ιούλιο του 2016. Ήδη από το 2015 θα πρέπει να υπάρξει μείωση για τις ε, τιμές λιανικής και θα ήθελα να υποστηρίξω τις τροπολογίες που γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση γιατί με αυτές οι εταιρείε θα εξοικονομήσουν χρήματα όχι εις βάρος άλλων, αλλά θα εξοικονομήσουν χρήματα επί τη βάση του αριθμού των πελατών που θα έχουν. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υποστηριχθεί αυτή η τροπολογία. Και να επανέλθω στο θέμα που αναφέρω συνεχώς, κάθε φορά πρέπει επιτέλους να καταργήσουμε αυτά τα διεθνή τέλη περιεγωγής που είναι πραγματικά ε, ε, παράλογα. Πρέπει να δώσουμε ένα τέλος σε αυτήν την κατάσταση. Η κυρία Στάιλερ. Θα είμαι σύντομη γιατί έχουν πολλά υποθεί από προλαλήσαντες συναδέλφους και νομίζω ότι πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση με τις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες. Ε, νομίζω η κατάργηση σταδιακή του, της περιεγωγής ε, με βρίσκει σύμφωνη. Την προτιμώ, αλλά πρέπει να έχουμε, να έχουμε εντωμεταξύ μεγαλύτερη προστασία μέσω ευελιξίας, καλύτερη τιμολόγηση. Νομίζω και η κυρία Βερνιό το είπε επίσης και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καλύτεροι ως προς την ενημέρωσή μας και ως προς τις υπηρεσίες. Νομίζω ότι η δυνατότητα αλλαγή συμβολέου είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι επιτέλους ε, έχει προχωρήσει. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά εδώ και πολλά χρόνια για αυτό το θέμα. Επιτέλους πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να υποστηρίξουμε τη βέλτιστη πρακτική όπου υπάρχει αυτή αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα των εμποδίων στην εσωτερική αγορά που παραμένουν. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για όλη τη δουλειά που έχει γίνει. Περιμένω τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αύριο βέβαια την ψηφοφορία μας. Ε, σε 119 ημέρες έχουμε εκλογές. Α, μετράτε τις ημέρες εγώ δεν τις μετράω με τόσο ζήλο. Yo creo que es un trabajo... Eh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά και κινείται προς αυτά που προστατέσαμε και υπερασπιστήκαμε στην Επιτροπή τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, η κυρία Μπάστος ε, έκανε έξοχη δουλειά και το έγγραφο είναι στο ύψος ε, αυτών που ήθελε ο εισηγητής και οφείλουμε και στην... και η δουλειά που έγινε είναι πάρα πολύ καλή, είναι έξοχη όσον αφορά τα αυτά που πρέπει να διευκρινιστούν. Νομίζω ότι θα γίνουν μέσω συζητήσεων συμφωνίες. Και θέλουμε τελικά το τελικό έγγραφο να είναι ακόμα καλύτερο από αυτό που έχουμε στη διάθεσή μας τώρα και συγχαρητήρια λοιπόν στον εισηγητή και στους ε, σκιώδεις ε, εισηγητέ. Αν δεν σας πειράζει θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες από πλευράς εισηγητού επί ενός σημείου. Νομίζω ότι από ό,τι κατάλαβα δεν θα αναφερθούμε στην περιαγωγή διότι δεν ενέπιπτε στις αρμοδιότητες της Επιτροπής αυτής. Εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας να θέσουμε τέρμα στον κατακαιρματισμό της αγοράς και να μειώσουμε το βάρος του καταναλωτού. Νομίζω ότι η περιαγωγή όσον αφορά αυτό το θέμα εμπίπτει τελικά σε αρμοδιότητα της Επιτροπής για τους λόγους που προανέφερα και θα έπρεπε να αναφέρεται στο τελικό κείμενο. Ήδη ε, υποβάλαμε ε, βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες λύσεις για την περιαγωγή και νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο σημαντικότατο κείμενο διότι έτσι οι μικρομεσές επιχειρήσει θα βοηθηθούν και οι καταναλωτές. Ίσως θα μπορούσε να μας διαφωτίσει περισσότερο ο εισηγητής επ' αυτού. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ο Άντωνι Βίλαν ίσως μπορεί να πει κάποια πράγματα, μέχρι έχουμε χρόνο. Και Σύντομα θα μπούμε και στο θέμα των ταξιδιών, πακέτων ταξιδιών. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βίλαν και μετά θα αναφερθώ στα θέματα της περιαγωγής. Ε, όταν θα συνοψίσω τη συζήτηση. Άντωνη Βίλαν, ευχαριστώ Πρόεδρε και συγκητά. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας συγχαίρουμε και εσάς και τους Κιώδης και την Επιτροπή σας. Ε, τάχιστος ο ρυθμός που ακολουθήσατε. Υπήρξε χρονική πίεση, ανταποκριθήκατε με επιδεξιότητα. Δεν στοιχηματίζω Οπότε θα προσπαθήσω να δω ποιες είναι οι πιθανότητες να σας πείσω εσάς και τους σκιώδεις σας το επόμενο 24 ώρα ότι βέλτιστο μέσο θα είναι η μέγιστη εναρμόνιση και σχετικός κανονισμός. Αλλά σημειώνω τις ε, απόψεις που εκφράσατε ξεκάθαρα το θετικότατον προσημείωση Συμβαστικές τροπολογίες είναι ο βαθμός στον οποίο η ουσία της προτάσεως Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προστασία του Ελικού Χρήστου έχει συμπεριληφθεί στην πρότασή σας. Πριν από λίγες εβδομάδες είχα μιλήσει στην Επιτροπή σας αναφερόμενος αυτό και είναι ευπρόσδεκτο ότι αυτή τη γραμμή και ευχαριστώ και τους Κιώδης για τη συνεισφορά τους στη σχετική. Βέβαια καλωσορίζουμε μεταξύ άλλων και αυτό που ζητάει η κυρία Βερνιό για το θέμα τερματισμού σε εξάμεινο. Θέμα προς διευκρίνηση. Για την προστασία του τελικού χρήστη εν γέννη. Είμαστε τελική ευθεία. Το είπε και η κυρία Μπάστος. Δύο σημεία πρέπει να προσέξουμε που μπορούν να βελτιωθούν στον διαθέσιμο χρόνο πριν την αυριανή ψηφοφορία. Ένα είναι αυτό που αναφέρατε, Πρόεδρε. Πώς καθορίζουμε τις ταχύτητες που αναφέρονται προσυμβασιακά και συμβασιακά και που αναγγέλλονται στον τελικό χρήστη. Χρειάζεται προσπάθεια για να μπορεί να εφαρμοστεί πράγματι για τους καταναλωτές. Η ελάχιστη αναμενόμενη ταχύτητα ε, δημιουργεί αμφισημίες όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής και επιβολής από τους καταναλωτές. Και το άλλο που ανέφερε η κυρία Βερνιό για διάρκεια συμβάσεων. Λοιπόν, για τη μεταφορά συμβάσεων, πώς μεταφέρεται το χρονικό όριο. Ίσως Πώς καλύπτουν οι συμβάσεις τα ενδεχόμενα κενά. Αυτό πρέπει να εξεταστεί. Μπορεί να το εξετάσουμε το επόμενο 24ωρο ή καθοδόν προς την Ολομέλεια και τη δουλειά που θα ακολουθήσει μετά στο Συμβούλιο για τη ρύθμιση λεπτομεριών. Για το ανοιχτό διαδίκτυο. Εάν σωστά αντιλαμβανόμαστε από το κείμενο, καλωσορίζουμε την πρόοδο για, την, για τον καλύτερο καθορισμό των, ειδικευμένων, των ειδικών υπηρεσιών όσον αφορά τη χωρητικότητα και τον αυστηρό έλεγχο. Για να αποφευθούν όμως αμφιβολίες πρέπει να γίνει η συμπλήρωση που προτείνει η κυρία Βερνιού. Πρόεδρε, και εμείς ανησυχούμε στο, για το εξής ότι οι εξειδικευμένες υπηρεσίες πρέπει να είναι συμπλήρωμα της ε, πρόσβασης στο διαδίκτυο και όχι υποκατάστατο. Χρειάζεται σαφής διατύπωση. Δεν θα πρέπει να εννοείται ότι όλοι οι πάροχοι των ειδικών αυτών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι και πάροχοι πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παρόλο που είναι στον τομέα παροχής περιεχομένου. Όσον αφορά τα θέματα που αφορούν περισσότερο την Ήτρε, με την οποία θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσει όπως είπατε, θέλουμε να δούμε σαφέστερη δέσμευση από ό,τι προβλέπεται στην πρόσβατη διατύπωση για ανολογική διαφανή και μη διακριτική διαχείριση της κυκλοφορίας και μέτρων και πρακτικών και όχι απλώς διαδικασιών. Και όπως είπε ο κύριος Κρόιτσμαν, ερχόμαστε στα κίνητρα για επενδύσεις. Πρέπει να αποφευθούν κενά όπου ίσως οδηγούν σε μόνιμη συμφόρηση και όχι προσωρινή και αυτό μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για να ε, ξεφύγουν οι διάφοροι πάροχοι από την ομοθεσία Και τέλος χρειαζόμαστε επιβολή των μέτρων. Άρα πρέπει να δούμε ουσιαστικές διατάξεις του άρθρου 23, το βασικό κείμενο, και τι γίνεται με τις διατάξεις περί εποπτείας και ελέγχου του άρθρου 24. Φαίνεται να είναι μακροσκελής ο κατάλογος. Μπορούμε να τα ρυθμίσουμε. Ούτως ώστε όλοι να είμαστε ικανοποιημένοι με τελική διατύπωση. Τέλος. Για τον αριθμό κλείσεως 112 που δεν συμπεριλαμβάνεται στην πρότασή μας. Ουδέν σχόλιον επί των λεπτομεριών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μελετήσει το θέμα δεόντως και θα έχει θέση ε, έγκαιρα πριν την Ολομέλεια. Αυτά και ευχαριστώ Πρόεδρε. Uh, thank you very Ευχαριστώ πολύ για τη θετική απόκριση υπερασπιστήκατε μέχρι τέλους τη θέση σας για τον κανονισμό. Θα δουλέψουμε επικοδομητικά για μια καλύτερη διατύπωση, όπως πιστεύουμε, υπέρ των καταναλωτών και θα δούμε και τον κανονισμό για την ανοιχτή πρόσβαση. Τον επόμενο μήνα θα γίνει περισσότερη δουλειά. Εγώ Προς το παρόν έκανα κάποιες προσθήκες ακόμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα υπάρξουν πολλές παραλλαγές γλωσσικές. Θα δούμε και με τους εισηγητές από την Επιτροπή Βιομηχανίας και την Επιτροπή Γιούρη. Τώρα, κάποια επιμέρους ζητήματα Συνεχώς υποστηρίζαμε το πακέτο για την περιαγωγή της Επιτροπής Βιομηχανίας και τα θέματα που αφορούν τους καταναλωτές και την ενημέρωση, ιδιαίτερα ενημερωτικά μηνύματα που παίρνουμε όλοι. Αυτά όμως δεν είναι προσυζήτηση αυτή τη στιγμή. Εγώ σε μεγάλο βαθμό υποστήριξα τη θέση του εισηγητή της Επιτροπής Βιομηχανίας που λέει ουσιαστικά ότι πρέπει να ε, καταργηθούν μέχρι το 2016 οι χρεώσεις για περιαγωγής. Δεν θέλουμε ενδιάμεσα μέτρα, δεν θέλουμε ε, ε, τίποτε, καμία χρέωση. Αυτός είναι ο στόχος. Βέβαια τώρα έχουμε μια ψήφο πρώτη, ψηφοφορία πρώτης ανάγνωσης και μετά θα πάει το θέμα για να το εξετάσουν τα κράτη-μέλη. Η ιδέα της αλλαγής της νομοθεσίας για την πειραγωγή ένα χρόνο πριν ε, λήξει δεν είναι ρεαλιστικό. Δεν διαφωνώ δηλαδή με ορισμένα από αυτά που λέτε, αλλά δεν είναι πρακτικά. Θα ξαναδώ κάποια ζητήματα όμως. Υπάρχουν ορισμένοι τομείς που δεν έχουν ε, ε, τύχει επεξεργασία στην Επιτροπή τη δική μας, αλλά την Επιτροπή Βιομηχανίας. Συνολικά περιμένω να υποστηρίξετε την πρόταση. Ευχαριστώ για τις συμβιβαστικέ. Θα μιλήσουμε για τις εξάμεινες συμβάσεις αύριο που νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική προϋπόθεση. Κάποιοι μπορούν να το έχουν ως προαιρετική. Αυτό θα ψηφιστεί ως προσθήκη αν θέλουν να το υποστηρίξουν και κάποιες άλλες διατυπώσεις θα είναι προσθήκες και θα δεχτώ την ψήφο της Επιτροπής πάνω σε αυτά. Και περιμένω να ε, συζητήσουμε και με την Επιτροπή Βιομηχανίας. Φαντάζομαι δεν έχουμε δει την πρόταση για την Ολομέλεια, αλλά αν στις 27 Φεβρουαρίου εγκρίνει η Επιτροπή Βιομηχανίας, μπορεί να πάμε για την Ολομέλεια του Απριλίου που θα είναι η τελευταία ευκαιρία. Καλό θα είναι να είστε παρόντες για να υποστηρίξετε τη θέση της Επιτροπής στην Ολομέλεια του Απριλίου, γιατί είναι πιθανό να γίνει αυτό. Ε, φροντίστε να είστε ελεύθεροι. Ευχαριστώ όλους πολύ. και ο κύριος Κρόιτσμαν, ε, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κρόιτσμαν, την ε, Νέσε, την, ε, τον Σεμπάστιαν, γιατί τις τελευταίες εβδομάδες δουλέψαμε μέχρι αργά για να προλάβουμε. Όλοι έκαναν πολύ καλή δουλειά, με υποστήριξαν και δεν θα τα κατάφερνα χωρίς εκείνους. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Πίσω από κάθε εισηγητή υπάρχει μια ισχυρή ομάδα και αυτό σίγουρα συνέβη εν προκειμένου. Τώρα, για τα ταξίδια Πρέπει να δούμε τις τροπολογίες εδώ για τα οργανωμένα ταξίδια. Ο Χάνς Πέτερ Μάιερ είναι εδώ, είναι ο εισηγητής. Λοιπόν, ας φύγουν όσοι δεν ενδιαφέρονται γι' αυτό, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε. Λοιπόν, εξέταση τροπολογιών. Είναι εδώ η εισηγητής ο Χάνς Πέτερ Μάιερ, το είπαμε. Από τους φιλελεύθερους κανείς, ο κύριος Κοφεράτη είναι εδώ για τους σοσιαλιστές, ε, ε κυρία Μακάρθη, κυρία Ζίντελ όλοι είναι σχεδόν, όλοι οι σχεδόν είναι εδώ. Κυρία Βανφρέντη, ποιος είναι εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριος Πέτρη. Oh, Mr. Matiak, is that right? Yeah. Okay. Anyway, we... Mr. Matiak will be speaking. Okay, all right. Well, thank you very much. Well, you're very welcome anyway. Uh, so, um, Hans Peter. Λοιπόν, Hans Peter. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, και αυτή η οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια και τους εξατομικευμένους διακανονισμούς μας φέρνει κάτω από χρονικές πιέσεις. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις και τους συνεργάτες τους. Συνολικά ήταν 435 οι τροπολογίες, πολλή δουλειά δηλαδή. Τις επόμενες μέρες θα συναντηθούμε με τους σκιώδεις και θα προσπαθήσουμε από όλες αυτές τις τροπολογίες να καταλήξουμε σε καλές συμβιβαστικές ιδιαίτερα προς το συμφέρον των καταναλωτών. Επειδή οι τροπολογίες είναι πολύ διαφορετικές, θέλω να αναφέρω μόνο τα σημαντικότερα σημεία σήμερα, για τα οποία μίλησα και με τους κοιόδης και πάνω στα οποία θέλω να επιτύχω συμβιβαστικές. Πρώτον, ο, βαθμός της εναρμόνισης. Όπως ανέφερα στην έκθεση, η διατύπωση που επέλεξα προέρχονται ε, κυριολεκτικά από την οδηγία για τους καταναλωτές. Θέλω η ευρωπαϊκή νομοθεσία να είναι όσο γίνεται πιο συνεκτική όταν έχουμε μια διατύπωση για το βαθμό της εναρμόνισης στην προστασία καταναλωτών, δεν πρέπει να επιλέγουμε και να εφευρίσκουμε συνεχώς καινούργιε διατυπώσεις ενώ κατ' ουσίαν εννοούμε το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν η διατύπωση είναι από την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Μετά τα κράτη-μέλη ε, μπορούν να έχουν ε, εθνικές διατάξεις εφόσον αυτές ε, ε, ρυθμίζονται σαφώς και καλύπτονται από την οδηγία. Εκεί που επιτρέπονται οι εξαιρέσεις, τα κράτη-μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν. Ο στόχος είναι κάθε καταναλωτής στο σύνολο της Ένωσης να γνωρίζει ποια δικαιώματα έχει. Ανεξάρτητα από το που θα κάνει την κράτηση, σε ποια χώρα, από πού θα κάνει την κράτηση, ποιος θα είναι ο ταξιδιωτικός προορισμός. Θέλουμε μια εσωτερική αγορά και οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς πρέπει να εναρμονιστούν ε, με όσο γίνεται λιγότερες εθνικές εξαιρέσεις. Και οι επιχειρήσεις πρέπει να ξέρουν ποια δικαιώματα έχουν σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί αν είμαστε σοβαροί με την ελεύθερη διακίνηση, ο καθένας από κάθε χώρα, μια επιχείρηση μπορεί να κάνει κρατήσεις στη Γερμανία, την Ισπανία και δεν πρέπει να ρωτάει κάθε φορά η επιχείρηση τι δικαιώματα υπάρχουν ε, σε κάθε περίπτωση ε, και για κάθε κράτηση. Όλα αυτά έχουν νόημα λοιπόν και ε, πρέπει να όλα να καταλήγουν στην καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Υπάρχουν λοιπόν και τροπολογίες για να ισχύσουν διαφορετικές ε, ρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει πάλι ότι κατακαιρματίζουμε την κυρωτική νομοθεσία σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει κάθε φορά να βλέπει κανείς τι ισχύει. Ενώ εγώ είμαι υπέρ των ενιαίων κανόνων σε μια ενιαία εσωτερική αγορά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις συμβάσεις online που πρέπει διασυνοριακά να λειτουργούν χωρίς πρόβλημα μέσω των κρατήσεων, γιατί καμιά φορά δεν ξέρουμε μια προσφορά από ποια χώρα προέρχεται και δεν με ενδιαφέρει αν η ε, προσφορά καθ' αυτή ε, είναι ενδιαφέρουσα. Αυτό τώρα για το βαθμό της εναρμόνισης. Το άλλο είναι το πεδίο εφαρμογής. Ε, υπάρχουν κάποιες προτάσεις στα επιχειρηματικά ταξίδια να εξαιρεθούν ολοσχερώς από το πεδίο εφαρμογής. Αυτό είναι δύσκολο για τους ελεύθερους ε, επαγγελματίες και τους μικροεπιχειρηματίες. Ε, σε κάθε νομοσχέδιο ε, εστιάζομαι στην κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικροεπιχειρηματιών. Αν κάποιος δικηγόρος, γιατρός, άλλος ελεύθερος επαγγελματίας πώς θα διαφοροποιήσει, θα είναι ιδιωτικό ταξίδι, θα είναι ε, επαγγελματικό, τι συνέπειες έχει κάθε φορά εάν το εξειδικεύει. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ευρύτερο το πεδίο εφαρμογής. Μεγάλοι επιχειρηματίες ε, πρέπει να εξεραθούν, δεν χρειάζονται την προστασία των συνήθων καταναλωτών, αλλά θα ήθελα πάνω σε αυτό να μου πούν τη γνώμη τους οι σκιώδεις συγητές, ούτως ώστε να οριοθετήσουμε σωστά, σωστά το πεδίο εφαρμογής. Τρίτο σημείο ε, ο ορισμός των οργανωμένων ταξιδιών, των εξατομικευμένων, ε, συνδεδεμένων ε, διακανονισμών ταξιδιωτικών. Δηλαδή, το κριτήριο διαχωρισμού έχει να κάνει με τον τρόπο της κράτησης και τον αριθμό των συμβάσεων ε, υπάρχει μία σύμβαση στα οργανωμένα ταξίδια πακέτο, στα εξατομικευμένα υπάρχουν περισσότερες συμβάσεις. Αυτό είναι ένα κριτήριο διαχωρισμού. Πρέπει να πω ότι η πλήρης διαγραφή των τελευταίων, των εξατομικευμένων, ε, δεν έχει νόημα, γιατί τότε ε, ε, χάνουμε το νόημα. Θα μπορούσαμε όμως να έχουμε συμβιβαστική λύση για καλύτερη οριοθέτηση και να καλύψουμε έτσι περισσότερες μορφές. Υπάρχουν προτάσεις για συμβιβαστικές, γιατί υπάρχουν ήδη ε, χρήσιμες ε, τροπολογίες που θα χρησιμεύσουν ως βάση για τις ε, συμβιβαστικές. Υπάρχουν τροπολογίες που προβλέπουν ένα, θέλουν το το στοιχείο της μεταφοράς και για, για τις δύο κατηγορίες για λόγους προστασίας των καταναλωτών δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό γιατί ε, οι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί με, ε, ε, με, όταν φτάνει κανείς στον προορισμό με δικά του μέσα αυτές δεν θα καλύπτονται και θα είναι μικρότερο, χαμηλότερο το επίπεδο ασφάλειας και προστασίας του καταναλωτή. Ε, πρέπει να το δούμε λοιπόν αυτό. Τέταρτο σημείο. μέχρι ποιο ποσοστό μπορούν να γίνονται αυξήσεις τιμών χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα υπαναχώρησης. Εδώ υπάρχουν διάφορες κλιμακούμενες προτάσεις, 3%, 5%, 7%, η Κομισιόν πρότεινε 10%. Θα το δούμε. Γιατί δεν υπάρχει ε, τώρα λύση ούτε υπάρχει πρόταση για λύση του τι θα συμβεί αν αυτά τα όρια 3, 5, 7% αν υπάρχει υπέρβαση αυτών των ορίων. Τι γίνεται τότε. Εγώ πρότεινα να μην υπάρχει μόνο δυνατότητα υπαναχώρησης αλλά και δυνατότητα από αντικατάστασης. Δηλαδή, ε, επίσης, ε, να υπάρχουν ρυθμίσεις για μειώσεις και όχι αυξήσεις τιμών επίσης, γιατί και αυτό μπορεί να συμβεί, να υπάρξει μείωση τιμής. Και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Ε, τι γίνεται αν βάλουμε ένα ποσοστό και γίνει υπέρβαση αυτού του ποσοστού. Θα πληρώσει ο επιχειρηματίας, η επιχείρηση, μπορεί κανείς να υπαναχωρήσει, ε, πώς θα γίνονται καταγγελίες κλπ. Ακόμα δεν έχω ε, ε, οριστική λύση. Τώρα, για την ευθύνη. Εδώ παίζει ρόλο ο αριθμός των διανυκτερεύσεων και το ύψος του αποκοπήν ποσού, δηλαδή που θα πληρωθεί. Ε, τι, πόσες διενυκτερεύσεις ε, θα εξασφαλίσει η επιχείρηση και ποιο είναι το ανώτατο όριο σε ευρώ. Εδώ ε, για τις πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις αεροπορικές εταιρείες. Αυτό θα αποφασιστεί το Φεβρουάριο. Νομίζω ότι κάτι παρόμοιο θα πρέπει να ισχύσει και εδώ. Δηλαδή καλό είναι να υπάρχει συμφωνία στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό εις ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις ε, και διανυκτερεύσεις. Τέλος, σχέση μεταξύ των οργανωτών και των ενδιάμεσων για ε, τα ταξίδια. Πρέπει να υπάρξει εδώ προστασία κατά της αφαιρεγγιότητας ε, και την ανάληψη ευθύνης. Πρέπει να είναι παρόμοια, ε, παρόμοιες οι λύσεις που θα προταθούν. Δεν έχουμε καταλήξει εις ό,τι αφορά τις επιπτώσεις που θα έχουν οι προβλέψεις. Οι οργανωτές και οι ενδιάμεση είναι δύο διαφορετικοί φορείς και εις ό,τι αφορά το μεγεθός τους έχουμε μικρούς ενδιάμεσους, έχουμε και μεγάλους, έχουμε ενδιάμεσους διαμεσολαβητές που είναι μικρομεσαίοι και δεν μπορούν να αναλάβουν ευθύνη, αλλιώς αν συνέβαινε αυτό θα έπρεπε να κλείσουν την επιχείρηση, άρα λοιπόν πρέπει εδώ να τα οριοθετήσουμε καλά. Αυτά είναι κάποια από τα σημαντικότερα σημεία που έχω εντοπίσει εγώ Όλοι νομίζω θα προσπαθήσουμε για να ε, επεξεργαστούμε καλή συμβιβαστική λύση. Ε, είναι, υπάρχουν χρονικές πιέσεις, γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν γρήγορα οι συναντήσεις των σκιωδών και πρέπει μετά από κάθε συνάντηση να, θα πρέπει να προσπαθούμε να συνοψίζουμε τα αποτελέσματα ε, της συζήτησης και να σας τα στέλνουμε. Η, χτες έγινε η ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή Τραν, θα αξιολογηθεί και αυτή και μετά θα προχωρήσουμε πιο γρήγορα νομίζω. Αλλά και οι συνεργάτες μας ε, ε, αντιμετωπίζουν μεγάλες πιέσεις. Αυτό είναι η συνέπεια των χρονικών πιέσεων και λόγω των επικείμενων ευρωεκλογών. Ευχαριστώ και με ενδιαφέρον θα περιμένω τις αντιδράσεις των αγαπητών συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Εκτιμούμε την ένταση των εργασιών και εγώ έχω τα ίδια προβλήματα με τις ανακοινώσεις. Είναι δυσχερέστατες οι συνθήκες στις οποίες εργαζόμεθα. Ο κ. Κονφεράτης, σαν εισηγητής, σαν σκιώδης εισηγητής του S&D. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε και για την πλήρη τοποθέτηση της έκθεσής του. Συμφωνώ Και αυτό διευκολύνει το έργο και των σκιωδών εισηγητών και, την, ε, και τις συμβαστικές. Θα περιοριστώ και εγώ, όπως και εκείνος, να αναφερθώ στα πιο ευαίσθητα σημεία κατά την απόψή μου και πιο περίπλοκα προς επίλυση ζητήματα που πρέπει να επιληθούν μέσω συμβιβασμών και οι συζητήσεις μεταξύ σκιωδών θα ρίξουν φως στις λεπτομέρειες. Δεν θα αναφερθώ τώρα σε λεπτομέρειες. Πρώτο πρόβλημα είναι της εναρμόνισης. Συμφωνώ ότι η αναφορά θα πρέπει να είναι της οδηγίας για την προστασία των καταναλωτών. Δεν έχω αντίρρηση. Όμως θα ήθελα να είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η εναρμόνιση είναι κοινή βάση. Είναι το, το, το, πάτωμα του, του σπιτιού και όχι η στέγη. Αν θέλουμε να υπάρχουν συμπληρωματικέ ε, προδιαγραφές για κάθε χώρα, θα πρέπει να έχω σαν στόχο τη βελτίωση της καταστάσεως για τον καταναλωτή και όχι το αντίθετο. Είναι θεμελιώδες να υπάρχει κάποια ομοιομορφία, αλλά μην εμποδίσουμε εκείνο που μπορεί ή θέλει να κάνει περισσότερα πράγματα, καλύτερα πράγματα. Η αρχή λοιπόν, κατά την άποψή μου, είναι αυτή. Μπορούμε να ετοιμάσουμε ένα σχετικό κειμένο για να εγγυηθούμε αυτή την υποθετική αλλά δυνατή βελτίωση μέσω αποφάσεων των κρατών μελών. Το πεδίο εφαρμογής είναι περιπλοκότατο ζήτημα, αντικειμενικά περιπλοκότατο. Πιστεύω όμως ότι θα ήταν χρήσιμο να μην αφαιρέσουμε τις ε, τουριστικές υπηρεσίες με βοήθεια που, ε, που αναφέρονται. Και αυτοί οι καταναλωτές πρέπει να προστατεύονται που χρειάζεται κάποια βοήθεια. Μιλάμε ότι υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι που χρειάζονται κάποια βοήθεια. Διαφορετικά αποκλεισμό αυτών των ανθρώπων θα θεωρηθεί σαν διάκριση. Νομίζω ότι το κείμενο, ένα κείμενο συμβιβαστικό μπορούμε να το επεξεργαστούμε, ούτω ώστε να καλύψουμε και αυτή την περίπτωση. Αυτούς τους χρήστες που χρειάζεται συνοδεία και να καλυφθούν οι ανάγκες τους. Για άλλα ζητήματα. Για προσυμβασιακή ενημέρωση. Τα δεσμευτικά χαρακτηριστικά της μεταφοράς των συμβάσεων. Αλλαγή τιμής κατά τη σύνευση της σύμβασης είναι σημαντικό να εργαστούμε με αυτό το πνεύμα με στόχο την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής βεβαιότητας όσον αφορά το σεβασμό της συμβάσεως και της καλύτερης δυνατής ενημέρωσης του καταναλωτού. Δεν θα πρέπει να θεωρείται ο καταναλωτής, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, σαν ανυπεράσπιστο παιδί, είναι ένα άτομο στο οποίο πρέπει να δίνονται όλα τα στοιχεία, να είναι ενήμερο και να κάνει τη σωστή επιλογή. Μπορεί να υπάρχει πληροφόρηση μέσα του δικτύου, αλλά είναι απαραίτητο κάποια φορά, κάποιες φορές, να δίδονται πληροφορίες στο χαρτί. Παλιές μέθοδοι ενημέρωσης, που δίνουν όμως τη βεβαιότητα αποφυγής απρόπτων για τον καταναλωτή. Πρέπει να βοηθήσουμε τον καταναλωτή με άλλα λόγια να έχει πλήρη επίγνωση των προσφερομένων και να αποφασίζει. Και πρέπει αυτό να καλύπτεται καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ό,τι σε εθνικό. Και να είναι δεσμευτική η ενημέρωση, να υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης. Στα νέα μέσα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και νέα μέσα πάντα με σκοπό την, να βοηθήσουμε τον καταναλωτή να επιλέγει. Το ανέφερε και ο συνάδελφος Ταραμπέλα αυτό. Να δίδονται ορατές ενδείξεις που θα αφορούν τον χαρακτήρα των προσφερωμένων πακέτων και των προσφερωμένων υπηρεσιών. Τι ούτω τρόπος τα πακέτα των ταξιδίων να αναφέρονται με ένα πράσινο σήμα και όταν δίδονται, παρέχονται υπηρεσίε με κάποια βοήθεια, να έχει διαφορετικό χρώμα, ένα σηματάκι με διαφορετικό χρώμα. Να μπορεί πιο εύκολα να βλέπει ο καταναλωτή, να ξέρει περί τίνο πρόκειται. Από την αρχή. Αυτές τις παρατηρήσεις έχω. Αυτά είναι τα πιο περίπλοκα ζητήματα. Στη συνεδρίαση των σκιωδών αν το θεωρεί χρήσιμο και ο εισηγητής για την, για την εργασία του, μπορούμε να ρυθμίσουμε τις λεπτομέρειες. Εγώ είμαι έτοιμος να δώσω λεπτομέρειες για τα θέματα τα οποία ανέφερα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χέλβικ δεν μπόρεσε να έρθει. Ε, για λογαριασμό της θα κάνω κάποια σχόλια σχετικά με το προ, ε, σχετικά με την πρόταση. Ε, γενικά είναι ίσοι οι κανόνες του παιχνιδιού έτσι, ε, χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις όμως στο κείμενο της Κομισιόν για το πεδίο εφαρμογής. Για παράδειγμα, ο κ. Χέλβιγκ έχει αμφιβολίες σε σχέση με τις διακανονισμούς συνδεδεμένους ε, ε, δεν πρέπει να υπόκεινται. Ε, σε ό,τι αφορά επίσης ε, άλλες εξαιρέσεις βοηθητικών υπηρεσιών γιατί για το επίπεδο της εναρμόνισης ο κ. Χέλβικ λέει ότι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν το ίδιο επίπεδο εναρμόνισης και όσο αυτό είναι δυνατόν. Συμφωνεί με την προσθήκη νέου άρθρου με βάση το 4α γιατί από την ε, ε, νομοθεσία προστασία των καταναλωτών. Θα πρέπει να δούμε τι χρειάζεται και είναι χρήσιμο για τους ταξιδιώτες πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Προσοχή να μην ε, κάνουμε σύγχυση μεταξύ προσυμβατικών και άλλων πληροφοριών, που οι τελευταίες είναι πιο εκτενές. Ναι, σας παρακαλώ, διακόπτει ο πρόεδρος. Μιλάτε λίγο πιο αργά για τη διερμηνία, παρακαλεί ο πρόεδρος. Μάλιστα, Μάλκολμ, ευχαριστώ ο κύριος Χέλβικ μπορεί να συμφωνήσει με κάποιες προτινόμενες αλλαγές, για παράδειγμα γλώσσες όπου ε, θα ε, αναφέρονται οι βασικές πληροφορίες. Ελπίζει όμως να μην υπερφορτωθούν οι επιχειρήσεις. Επίσης, η ευθύνη για την παροχή προσυμβατικών πληροφοριών. Αυτή πρέπει να είναι ευθύνη των οργανωτών ή του λιανοπολιτή, αν το πακέτο το πουλήσει ένας λιανοπολιτής. Όπως ο εισηγητής και άλλοι συνάδελφοι, ε, ο συνάδελφος Χέλβικ στηρίζει την ιδέα να έχουν το δικαίωμα οι ταξιδιώτες ε, να ακυρώνουν χωρίς χρέωση το πακέτο σε περίπτωση αλλαγής στην τιμή πάνω από 10% και να υπάρχει υποχρέωση να παρέχονται σαφείς πληροφορίες για τέτοιου είδους αλλαγές τουλάχιστον 20 μέρες πριν από την έναρξη του ταξιδίου, του πακέτου. Επίσης θεωρεί ότι όταν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στη σύμβαση, ο ταξιδιώτης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποδεχτεί τις αλλαγές, να ακυρώσει χωρίς χρέωση το πακέτο ή να δεχτεί ισοδύναμο πακέτο που θα του προτείνει ο οργανωτής. Ο συνάδελφός μου δεν είναι πεπισμένος ε, για την ανάγκη να υπάρχει περίοδος υπαναχώρησης ε, για εξαποστάσεως ε, συμβάσεις γιατί αυτές συνάπτονται μετά από αίτημα του καταναλωτή. Γι' αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Για την ευθύνη θέλει να περιορίζεται η ευθύνη ε, στον οργανωτή για τη λειτουργία του πακέτου. Σε περίπτωση όπου ο οργανωτής δεν μπορεί να διακανονίσει την επιστροφή, να ρυθμίσει την ε, επιστροφή των ταξιδιωτών, ο κ. Σέλβιγκ θα πρέπει να ε, θέλει να συζητηθεί το ύψος της αποζημίωσης, του κόστους που θα καλύψει ο οργανωτής, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, λέει, για να μην το παρακάνουμε, γιατί αυτό θα επηρεάσει πολύ αρνητικά τις μικρές επιχειρήσεις, τα μικρά ταξιδιωτικά γραφεία και μου φαίνεται ότι ο κύριος Μάιερ το ίδιο είπε πριν από λίγη ώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρούλε. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για τις προσπάθειες που έκανε μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα να διευκρινίσει θέματα. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι 438 τροπολογίες και η διαφορετικότητά τους, γιατί είναι και πολύ διαφορετικές ε, στο περιεχόμενο. Η τροπολογία δείχνει ότι δεν έχει προχωρήσει η συζήτηση ακόμα πολύ. Καλύτερα να είχαμε αρχίσει με ένα ψήφισμα και να μην αρχίζαμε όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά το είχαμε συμφωνήσει τέλος πάντων. Τώρα πρέπει να δούμε τι καλύτερο μπορεί να βγει από αυτή την ιστορία. Ε, εγώ πρέπει να πω ότι ε, εστίασα την προσοχή μου σε συγκεκριμένες τροπολογίες αλλά χρειάζεται κι άλλη συζήτηση διότι ακόμα υπάρχουν πολλές ασάφειες βαθμός ε, της εναρμόνισης. Έχουμε πρόβλημα με τη μέγιστη εναρμόνιση που επιδιώκεται στην οδηγία προστασίας καταναλωτών γιατί σε κάποιους τομείς ε, δεν υπάρχει ε, ομοιομορφία και έχουμε αμφιβολία αν μπορεί να υπάρξει μέγιστη εναρμόνιση, πλήρης εναρμόνιση. Σημαντικό είναι επίσης να ορίσουμε και αυτό είναι πιο σημαντικό το πεδίο εφαρμογής. Επαγγελματικά ταξίδια δεν επικεντρώνω εκεί την προσοχή μου. Πρέπει να δούμε τι δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας ε, μιλάμε για ε, οργανωμένα, ε, συνδεδεμένα, αλλά υπάρχουν και πολλοί συνδυασμοί που κάποιοι φτιάχνουν μόνοι τους προσθέτοντας κάποια στοιχεία και εκεί δεν υπάρχει διασφάλιση και αναλαμβάνουν οι ίδιοι το ρίσκο. Και αυτό θα πρέπει να είναι δυνατό να γίνεται. Έχω την εντύπωση, βλέποντας κάποιες τροπολογίες, ότι αυτό πάει να αποκλειστεί ούτως ώστε κάθε ταξίδι στο μέλλον να εμπίπτει αυτή, στο πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Ε, ανησυχώ λοιπόν γιατί είναι πολλές τροπολογίες αυτές. Γιατί ε, δεν νομίζω ότι ε, θέλουν μείωση της προστασίας. Το σημαντικό είναι όμως να υπάρχει διαφάνεια. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη, ποιος έχει την ευθύνη γιατί. Ε, αλλά θα πρέπει να είναι δυνατόν αν κάποιος θέλει να φτιάξει ένα πακέτο ταξιδίου μόνος του να μην είναι υποχρεωμένος να ε, κάνει έναν εξατομικευμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό. Επίσης θα πρέπει να δούμε και τη σχέση με τα δικαιώματα, ε, με την οδηγία για τα δικαιώματα των ταξιδιωτών. Μπορούμε εδώ να βρούμε ε, συμβιβαστικέ λύσεις πιο εύκολα. Το βασικό είναι να ορίσουμε το πεδίο εφαρμογής, τι στην οδηγία, τι δεν εμπίπτει και ποιες είναι οι επιπτώσεις. Uh, thank you very much, Mrs. Κύριε Μακλάρτιν, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες, ελπίζοντας να ενισχύσω το κείμενο σε βασικά ζητήματα της περιόρισα και σε αυτό θα περιοριστώ και σήμερα όπως είπε και ο κύριος Μάιερ, ε, πρέπει να υποφελούνται από την οδηγία αυτή κυρίως οι κατανάλωτες και δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις. Βέβαια καταλαβαίνω τα προβλήματα που ε, εντόπισε και ο κύριος ε, Μάιερ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες που λένε ότι εκτός από την εταιρική επωνυμία θα μπορούσαν να καλύπτονται και από αυτή την οδηγία. Ε, όσον αφορά τώρα τις ε, εξατομικευμένες υπηρεσίες, νομίζω ότι πρέπει να καθορίσουμε τι θα πει ε, ιστότοπο σύνδεσης, δηλαδή που σε πάει σε ένα άλλο ιστότοπο για να κάνεις μία άλλη κράτηση. Όσον αφορά τώρα τους επιβάτες, πρόκειται για μία οδηγία για ταξιδιωτικέ υπηρεσίες. Προφανώς θα περιλαμβάνει κάποια πράγματα για του επιβάτες. Αν αναφερέστε στις ε, προσωπικά ταξίδια, για παράδειγμα κάποιο πηγαίνει με ένα λεωφορείο να μείνει σε ένα ε, ξενοδοχείο και να πάει θέατρο, αν κάποιο αποφασίσει να πάει ε, στο αν κάποιο αποφασίσει να μην κάνει όλο το πακέτο, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα πρέπει να χρήζει περαιτέρω κάλεψης από την εν λόγω εταιρεία. Ε, βέβαια οι καταναλωτές ε, πρέπει να γνωρίζουν 100% για το κατά πόσο πρόκειται για τη μία ή την άλλη μορφή ε, ταξιδίου και αν θέλουν πακέτα ταξιδίων να να κλείσουν πρέπει να καταλαβαίνουν το επίπεδο της προστασίας που έχουν ή δεν έχουν. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να είναι σαφές αυτό πριν, πριν από την πληρωμή του εν λόγω πακέτου. Επίσης πρέπει να επικεντρωνόμαστε περισσότερο στο πώς ε, τι διατίθεται στους ε, καταναλωτές και στην αγορά αυτό το πακέτο, ειδικότερα για το συγκεκριμένο κομμάτι του ταξιδιού που συμπεριλαμβάνεται ή όχι, αν υπάρχουν πακέτα με επιπλέον ε, παροχές που δεν αποτελούν όμω την ουσία, το σημαντικότερο τμήμα του πακέτου. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν πώς γίνεται η διαφήμιση στον καταναλωτή και κυρίως ε, στα έντυπα τα διαφημιστικά φυλάδια. Ίσως αν γίνει πάρα πολύ εναρμόνιση να μην υπάρχουν πια τα ωφέλη που έχουμε σήμερα. Οπότε πρέπει να στοχεύσουμε την εναρμόνιση ώστε οι καταναλωτές ε, να μην ε, βλάπτονται. Σε σχέση τώρα με τις τροπολογίες που έχουν υποβάλει κάποιοι συνάδελφοι, έχω κάποιες ανησυχίες. Για παράδειγμα, η, το αυτόματο δικαίωμα υπαναχώρησης από ένα ταξιδιωτικό συμβόλαιο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο και μιλάω τώρα για τις κρατήσεις τελευταία στιγμή σε ξενοδοχεία που είναι τεράστιο βάρος ε, για ε, τις ε, επιχειρήσεις αν ο πελάτης τους έχει τη δυνατότητα αυτόματης υπαναχώρησης από το συμβόλαιο. Τώρα τα συγκεκριμένα μοντέλα ε, κράτησης ε, ταξιδίων ε, τα οποία αναφέρουν, αναφέρουν οι συγκεκριμένες οδηγίες δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αποτελούν τμήμα της οδηγίας για τις τροπολογίες 151 και 152 αφορούν υπηρεσίες που αφορούν κρατήσεις που έχουν μια περίοδο ε, ανάκλησης 24 ωρών. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε με λίγο περισσότερη προσοχή αυτή, αυτό. Και στην 388 ε, τροπολογία ο λιανοπολιτής και ο οργανωτής ε, πρέπει να αναλάβει την ευθύνη αφαιρεγγιότητας. Δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να υπάρχει αυτή η διπλή προστασία και αν είναι απαραίτητη ή ο ένας ή ο άλλος θα έπρεπε να αναλαμβάνει την ευθύνη των διατάξεων αυτών. Αλλά ούτως ή άλλως θα τα συζητήσουμε αυτά ε, στις συναντήσεις με τους σκιώδεις εισηγητές μας σε μεταγενέστερο στάδιο. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε. Θέλουμε να είναι ποιοτικό το κείμενο που θα προκύψει. Έχουμε πάρα πολλά ακόμη να κάνουμε σε σχέση με τα επίπεδα εναρμόνισης αλλά θα ήθελα να το συζητήσω και με τον κύριο Μάιερ και με τους υπόλοιπους κοιόδης συζητητές το απόγευμα, για να μπορέσει να προκύψει κάτι το οποίο θα είναι σαφές, πολύτιμο και για τους καταναλωτές και για τους ε, επιχειρηματίες. Ευχαριστώ. Thank you very much to all the... Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους κοιόδης συζητητές για, αυτές τις, ε, για αυτά τα πολύ επικοδομητικά ε, σχόλια. Η κυρία Στάιλερ θέλει να πάρει το λόγο. Θέλει κανείς άλλος? Κυρία Στάιλερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ τον ε, ε, εισηγητή και τους Σκιώδης. Νομίζω ότι μπορώ να συμφωνήσω με όλους όσους είπαν για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Ε, θα ήθελα να δω τις συμβαστικές λύσεις που θα προτείνει ο κύριος Μάιερ. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τελικά. Η κυρία Ριούλε το είπε. Το θέμα είναι ποιο έχει την ευθύνη γιατί και πώ εξασφαλίζουμε την προστασία των καταναλωτών σε όλη αυτή τη διαδικασία, να καταλαβαίνουν πολύ καλά ποια είναι τα δικαιώματά του. Νομίζω ότι την ώρα υπάρχουν πολλά ανεπίλητα, ε, αναπάντητα ερωτήματα ε, και φαίνεται να υπάρχουν κάποιες φαιές ζώνες οι οποίες αποδυναμώνουν τα, τα δικαιώματα των καταναλωτών, των καταναλωτών γιατί δίνουν παραθυράκια είναι ένα συμβιβαστικό πακέτο και η σκληρή δουλειά των σκιωδών ε, σήμερα τα απόγευμα συνάντησή τους θα είναι κρίσιμη. Για το χρονοδιάγραμμα, ξέρω ότι οι συμβαστικέ τροπολογίε θα τι λάβουμε, ελπίζω, σε όλε τι χώρε, σε όλε τι γλώσσε το συντομότερο δυνατόν. Αυτή τη στιγμή συμφωνήσουν οι σκιώδει ε, οι εισηγητέ. Αλλά επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και επειδή οι συνεδριάσεις μας ε, είναι όλο και ε, λιγότερο συχνές. Θα τα καταφέρουμε μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής μας θητείας να ε, ολοκληρωθεί αυτό το ζήτημα. Με απασχολεί λίγο πιο πολύ το χρονοδιάγραμμα. Μήπως θα μπορούσε ο εισηγητής ή ο πρόεδρος να μας πει κάτι περισσότερο από αυτό. καλώς. Εν τη αυτή περίπτωση, αν συμφωνεί ο κύριος Μάιερ, θα προχωρήσουμε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάτια να σχολιάσει και μετά ο συγκεκριτής θα ξαναπάρει το λόγο. Έχετε το λόγο, κύριε Μάτιακ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να σχολιάσω όλες τις τροπολογίες. Δεν έχουμε χρόνο. Άρα δεν ενδεικνύεται. Ευχαριστώ τον εισηγητή και όλα τα μέλη της Επιτροπής σας εξετάσατε διεξοδικότατα το θέμα παρά την έλλειψη χρόνου. Όπως προαναφέραμε, οι πρώτες Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν καρπός διεξοδικότατων συζητήσεων και διαβουλεύσεων Είναι πολύ ισορροπημένη λύση. Είναι δυνατές με βελτιώσει σε κάποιους τομείς. Η βασική αρχιτεκτονική ιδέα της προτάσεως και το περιεχόμενο πρέπει να παραμείνουν έχουν. Συμπεραμονμόνησης της διάκρισης μεταξύ πακέτων και εξατομικευμένης ρύθμισης. Ήταν πολύ σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια να ξέρουν οι καταναλωτές ποιο ταξιδιωτικό προϊόν αγοράζουν. Η αδίποτε πρόταση ενισχύει τη διαφάνεια ευπρόσδεκτη. Γνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι πρέπει να δίδεται η σωστή ενημέρωση τη σωστή στιγμή. Δεν είναι ο όγκος που παίζει ρόλο των πληροφοριών. Σχετικά με αυτό προβληματιζόμαστε όσον αφορά προτάσεις περί χρώματος ετικετοθεσίας για ταξιδιωτικά πακέτα, κάποιου σήματος. Πριν εγκριθεί η πρόταση, αναθέσαμε μία μελέτη. Τα πορίσματά της ήταν μάλλον αρνητικά και αποθαρρυντικά περί αυτού. Σημαντικότερη είναι η θετική και αρνητική σαφής ενημέρωση. Να μην αγοράζει κανείς ένα πακέτο και να κάνει κρατήσεις εάν δεν είναι ενήμερος. Αυτές είναι πιο χρήσιμες οι πληροφορίες για τον καταναλωτή. Από ότι χρωματικοί κώδικες, κάποιο σήμα, κάποια ετικητοθεσία, οποιασδήποτε μορφής. Το επίπεδο εναρμόνισης. Εν συντομία υποστηρίζω τα όσα ανέφερε ο εισηγητής. μια, αν ακολουθήσουμε προσέγγιση εστιασμένης ή ελάχιστης εναρμόνισης και έτσι τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν περί των σημαντικών αλλαγών του νομικού πλαισιού, εάν γίνει αυτό θα αγνοεί τους στόχους της εσωτερικής αγοράς που περιέχονται στην πρότασή μας. Και δεν θα λάβουμε υπόψη την ψηφιακή διάσταση της πρότασης να μην λησμονούμε ότι σε μεγάλο βαθμό αναφερόμεθα σε υπηρεσίες μέσω διαδικτύου που παρέχονται online, διασυνοριακά. Τέλος, ευθύνες. Υπάρχουν διάφορες ανησυχίες που κρύβονται πίσω από διάφορες σχετικές ιδέες. Όμως μέχρι τώρα δεν πιστήκαμε ότι μία απόκληση από τη δική μας πρόταση θα ήταν επωφελής για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Προσεκτικά μάλιστα. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα σημεία. Σας εύχομαι καλή τύχη για να καταλήξετε στους βέλτιστους δυνατούς ε, στις βέλτιστες δυνατές συνενετικές λύσεις που θα είναι επωφελείς προς τους ε, καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο Hans ε, Peter Mayer έχει το λόγο για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους ε, που εξέφρασαν σύντομα τη γνώμη τους. Τα απόγευμα θα έχουμε την πρώτη συνάντηση των σκιωδών και θα εξεργαστούμε σε μεγαλύτερο βάθος κάποια πράγματα. Για τα χρώματα υπάρχουν μερικοί που δεν τα αναγνωρίζουν. Αν ας πούμε είναι πράσινο ένα πακέτο, ε, δεν θα το αναγνωρίσουν αυτοί που δεν βλέπουν τα χρώματα. Ε, θα θεωρήσουν ότι αυτό είναι ένα οποιοδήποτε άλλο ταξίδι. Ε, χρειάζεται λύση εδώ. Βέβαια για άλλους είναι καλή λύση τα χρώματα. Τώρα, ποιος καταναλωτής γνωρίζει ε, το ποια συγκεκριμένα δικαιώματα του παρέχει για παράδειγμα ένα ε, οργανωμένο ταξίδι. Πρέπει να δούμε πώς θα τα παρουσιάσουμε. Ο συνήθις ε, καταναλωτής πηγαίνει στο διαδίκτυο, κάνει την κράτησή του. Ε, πρέπει λοιπόν να βρούμε σωστό τρόπο για να έχει προστασία και αν δεν θέλει, όπως λέει και η κυρία Ρουλή, αν θέλει να αναλάβει ένα ρίσκο, γιατί εμείς θα πρέπει να επιμένουμε για το αντίθετο. Αυτό έχει να κάνει με την παροχή συμβουλών που έχει. Ε, δηλαδή, όπως λέμε, γιατί μου θυμώνεις, ε, εγώ δεν σου ε, παρήχα καμιά βοήθεια. Πάντως ε, ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να υποβάλουμε μια καλή συμβιβαστική πρόταση. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ για σας, εσάς και την ομάδα σας για τη δουλειά που κάνατε. Περιορισμένο χρονοδιάγραμμα, σημαντικότατο θέμα. Πληρέστατη γνωμοδότησή μας για το χρονοδιάγραμμα. Έχουν οργανωθεί διάφορες συναντήσεις. 11, μάλλον 10 Φεβρουαρίου συζητούμε τις συμβαστικές. Ψηφοφορία 11 Φεβρουαρίου και για... θα κινηθούμε για έγκριση στην Ολομέλεια του Μαρτίου. 10 Φεβρουαρίου. Συζήτηση συμβιβαστικών. 11 Φεβρουαρίου ψηφοφορία στην ΙΜΚΟ και πάμε μετά στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Καλώς. Ωραία. Τελευταίο σημείο προστασία καταναλωτών ε, όσον αφορά τις κοινοφελείς υπηρεσίες. Ο κύριος Χολτσάινερ είναι ο εισηγητής. Σας δίνω το λόγο για τις συμβαστικές. Η κυρία Γκέλπιρτς για το ΕΛΚ. Ο κύριος Σμιτ δεν είναι εδώ, ίσως να έρθει όμως. Η κυρία Ρούλε είναι εδώ και εγώ είμαι εδώ. Ο κύριος Χάντες δεν είναι εδώ έχετε αρκετούς σκιώδεις, οπότε μπορείτε ε, να ξεκινήσετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στον πρώτο γύρο τον Νοέμβριο κάναμε μια πολύ ζωντανή συζήτηση ε, που αφορούσε και το περιεχόμενο και τον, το πεδίο εφαρμογής της έκθεσης πρωτοβουλίας. Τονίζω ότι σε αυτό το τομέα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα κράτη-μέλη υπάρχουν διαφορές ως προς, την, προς τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, και πολλές φορές οι διαφορές αυτές που υπάρχουν οδηγούν σε σύγχυση μεγάλη. Και σίγουρα δεν διευκολύνει η κατάσταση αυτή την συζήτηση. Αντίθετα όμως οι υπηρεσίες κοινή ωφέλειας είναι ένα συνήθις ε, ε, ορισμός, ένας ε, όρος συνήθισε, οπότε πρέπει να μας απασχολήσει. Εγώ προσπάθησα να περιορίσω λίγο το εύρος της έκθεσης και να εστιάσω στις υπηρεσίες κοινή ωφέλεια μέσα από το πρίσμα του καταναλωτή και έτσι να κάνω συστάσεις για να βελτιωθεί η προστασία του καταναλωτή ως έχει σήμερα. Η έκθεση έχει υποδιαιρείται σε τέσσερις τομείς που είχαν απελευθερωθεί στο παρελθόν και ενσωματώθηκαν στην ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, συγκοινωνίες και ταχυδρομικές υπηρεσίες είχαν ενσωματωθεί στην ενιαία αγορά. Σε αυτούς περιορίστηκα. Βέβαια μπορεί κανείς να πει ότι ενδεχομένως και άλλοι τομείς θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν. Μετά την πρώτη συζήτηση ε, συνάντηση και συζήτηση για τις τροπολογίες κατάλαβα ε, πολύ περισσότερο από ό,τι όταν έκανα το πρώτο σχέδιο ότι δεν θα συγκεντρωθεί πλειοψηφία και δεν υπάρχει ενδιαφέρον για συμπληρωματικές, για πρόσθετες νέες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Δεν ζητάει κανείς κάτι τέτοιο. Οπότε έπρεπε να περιοριστώ στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και τις δυνατότητες που προβλέπονται εκεί. Τα τελευταία χρόνια μέσα από πολλά νομοθετικά μέτρα ε, βελτιώθηκε η προστασία των καταναλωτών. Παράλληλα όμως υπάρχουν ακόμα δυνατότητες και ανάγκες στα πλαίσια του υφισταμένου νομοθετικού πλαισίου για βελτιώσεις και νομίζω ότι αυτή είναι και η προσέγγιση που θα μπορούσε να συγκεντρώσει τη σύμφωνη γνώμη όλων. Οι αντιδράσεις στις τροπολογίες συνολικά ήταν επικοδομητικές, ε, εντόπισαν προβλήματα και ήταν πολλές, ήταν 156 συνολικά οι τροπολογίες που περιείχαν επικοδομητικές προτάσεις. Εγώ προσπάθησα να τις συνοψίσω, να τις συμπτύξω και να καταλήξω σε 19 συμβιβαστικές. Εδώ υπάρχει μια νέα παραλα... εκδοχή η οποία ετοιμάστηκε χθες μόλις που λαμβάνει υπόψη και τη συζήτηση που έγινε στην πρώτη συνάντηση των σκιωδών στο Στρασβούργο, όπου εκφράστηκαν κάποιες έντονες επιφυλάξεις ότι δηλαδή δεν πρέπει που δεν είναι να επιχειρήσουμε να δημιουργήσουμε καινούργιες αρμοδιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Ε, αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να συζητήσουμε ε, την τελευταία ε, εκδοχή από 21 Ιανουαρίου, από 19 Ιανουαρίου. Προσπαθώ να ε, ενισχύσω το θέμα της ενημέρωσης των καταναλωτών, πτυχές προστασίας, ρυθμίσεις για καταναλωτές ε, που χρειάζονται ιδιαίτερη μεταχείριση, ευάλωτες ομάδες, μεγαλύτερη συγκρισιμότητα ε, των παρόχων ενέργειας, ε, να δούμε επίσης και το ζήτημα της ενεργειακής παινίας, την αλλαγή του παρόχου, το smart metering, Σημαντικό είναι να δούμε και την αποτελεσματικότητα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, τη διαθεσιμότητα ε, αυτών των υπηρεσιών. Οπότε συνολικά έχω τις συμβιβαστικές τροπολογίες, κάποιες ε, απόψεις μου πολιτικές ε, τις απέσυρα και προσπάθησα να βρω έναν κοινό παρονομαστή μέσα από τις τροπολογίες. Το σχέδιο έχει κατατεθεί. Νομίζω ότι είναι δυνατόν επ' αυτής της βάσεως να καταλήξουμε σε κοινή θέση. Στάλησαν ε, στους σκιώδεις τα κείμενα στην τελευταία συνάντηση των σκιωδών δεν προλάβαμε να συζητήσουμε όλες τις τροποποιήσεις Λοιπόν, μπορούν να δουν η επόμενη, στις 30 Ιανουαρίου θα γίνει η επόμενη συνάντηση των σκιωδών για να συνεχίσουμε την επεξεργασία των τροπολογιών και έχουν σταλεί τα απαραίτητα έγγραφα ε, στη γραμματεία. Έτσι θα μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μας όλες τις απόψεις. Και φαντάζομαι ότι θα καταφέρουμε να επεξεργαστούμε κοινή θέση η οποία γενικότερα θα απηχεί τις συζητήσεις που έγιναν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία ε, Καλοπέλτς. Θα ήθελα και εγώ να παρουσιάσω την άποψή μου σε σχέση με τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Ε, εκπροσωπώ τον συνάδελφο Η διαφορά ήταν η ανάγκη νέων κοινών κανόνες παρά το γεγονός ότι υπήρξαν αλλαγές ε, δεν άλλαξε η βασική μου άποψη. Κατά τη γνώμη μου, οι νέοι δασμευτικοί κανόνες δεν ε, είναι απαραίτητοι, γιατί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι παρκές. Θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποτέ δεν προσπάθησε να δημιουργηθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο εναρμονισμένο για τις υπηρεσίες κοινή ωφέλεια, ε, γιατί είναι εθνική αρμοδιότητα και ευθύνη. Θα ήθελα λοιπόν να γίνει διαγραφή της αναφοράς στους κοινούς δεσμευτικούς κανόνες. Σκοπό έχω τα θεμελιώδη δικαιώματα να τα ενισχύσω διότι υπάρχουν και οι αρχές της ε, επικουρικότητας και της αναλογικότητας, ώστε να μην υπάρχει διπλή δουλειά και νομικές αντιφάσεις. Θα ήθελα επίσης να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για τους ε, για τον τομέα της ενέργειας, για παράδειγμα, ακόμα και καταναλωτικές οργανώσεις ε, ε, δεν θέλουν τόσο, ιδιαίτερη, τόσο έντονη παρέμβαση που μπορεί να ε, καταπατεί την εθνική αρμοδιότητα. Πρέπει να δούμε πού υπάρχουν κενά και να, να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικέ προκλήσεις. Αλλά δεν μπορώ να αποδεχθώ την αναφορά στις πρόσφατες μελέτες ε, για τους ευφυείς μετρητές, γιατί κάποιοι εξοικονομούν αλλά κάποιοι άλλοι όχι. Νομίζω ότι κάποια στοιχεία είναι αντιφατικά και κατά τη γνώμη μου δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε αυτά. Είμαι πεπισμένη ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της ε, οδηγίας ε, ε, για την ενέργεια δίνει τη δυνατότητα και στο, στα αυτοκίνητα να μειώσουν την κατανάλωσή τους. Νομίζω ότι γενικώ ο ενεργειακός τομέας αναφέρεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο πλαίσιο του κειμένου αυτού. Δεν χρειάζεται να αναφέρεται τόσο. Όσον αφορά τώρα τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, στο συμβιβασμό 17, για παράδειγμα, βλέπω μία αντίφαση μεταξύ την αύξηση της ποιότητας της υπηρεσίας και της εξοικονόμησης, κατά τη γνώμη μου. Πιο ποιοτικέ υπηρεσίες δεν σημαίνει υποχρεωτικά εξοικονόμηση χρημάτων στην περίπτωση αυτή. Απέστειλα την άποψή μου στον εισηγητή την περασμένη Παρασκευή. Ε, δυστυχώς ε, δεν έλαβε υπόψη τα σχόλιά μου σε σημαντικό βαθμό ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τον αναθεωρημένο, ε, τις αναθεωρημένες συμβιβαστικές ε, από, ε, απόψεις για την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Γκάλπεστ. Ο κύριος Μάντες εκ μέρους του κυρίου Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του συναδέλφου, αλλά μου έδωσε ένα σημείωμα να το διαβάσω βεβαίως και όπως ξέρετε πάντοτε βοηθώ τους φίλους. Ευχαριστεί λοιπόν τον εισηγητή για το συμβιβαστικό του πνεύμα και λέει ότι είναι, ένα πάρα πολύ, είναι πολύ πολιτική έκθεση ή πιστεύει κανεί ότι η πιστευει κανεις οτι Ένωση πρέπει να εισαγάγει νέους κανόνε για τι ε, υπηρεσίε κοινή ωφέλεια, είτε διαφωνεί. Δεν συμφωνεί με την εισαγωγή κανόνων προς αυτή την κατεύθυνση. Επίση, ο κύριο Σμιτ πιστεύει ότι οι ευάλωτοι καταναλωτέ, ο όρος αυτός, θα πρέπει να χρησιμοποιείται προσεκτικά, γιατί ο στόχο τη καταναλωτική πολιτική Ένωση είναι να ενδυναμώσει όλου του καταναλωτέ να κάνουν, ε, γνώ, να κάνουν εν γνώση τους επιλογές. Αν όλοι οι καταναλωτές θεωρούνται ευάλωτοι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι είναι αυτοί που χρειάζονται επιπλέον βοήθεια. Ευχαριστή λοιπόν τον εισηγητή για, την, για τις προσπάθειές τους. Αυτά εκ μέρου του κύριου Σμιτ. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομη ε, τοποθέτηση, αλλά χρήσιμη. Κυρία Ρουλέ. Ευχαριστώ τον εισηγητή που έδειξε πολύ μεγάλο συμβιβαστικό πνεύμα γιατί οι απόψεις στην Επιτροπή διήστανται εδώ, αποκλίνουν και χαίρομαι που δεν ζητάει κι άλλες οριζόντιες ε, ρυθμίσεις. Στις λεπτομέρειες εξακολουθώ να έχω κάποιες δυσκολίες γιατί οι τομείς αυτοί δεν ρυθμίζονται σε τομεακές ε, οδηγίες και είναι και πολύ διαφορετικοί οι τομείς μεταξύ τους με ελάχιστες ομοιότητες οπότε δεν υπάρχουν καθόλου σχεδόν οριζόντιες προτάσεις πρέπει Επίσης, ε, να, η συμβιβαστική 8 είναι πολύ προβληματική, για παράδειγμα, γιατί προβλέπει ότι ιδιαίτερα ευάλωτοι καταναλωτές θα πρέπει να απαλλάσσονται από χρεώσει. Δηλαδή θα πρέπει να προβλέπουμε για εξοικονόμηση ή μείωση ή διαγραφή του κόστους της χρέωσης για αυτούς. Πολύ προβληματικό θεωρώ, γιατί είτε μιλάμε για την ενέργεια, για τα ταχυδρομεία, για τις συγκοινωνίες, κάθε φορά υπάρχουν διαφορές. Υπάρχουν τομείς που έχουν τοπική εμβέλεια, όπως οι δημόσιες συγκοινωνίες, υπάρχουν άλλοι κεντρικές υπηρεσίες στα κράτη-μέλη και Ανάλογα με αυτό θα πρέπει και οι προσφορές και οι επιπτώσεις να είναι διαφορετικές. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι όλος αυτός ο τομέας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα από τομεακές οδηγίες. Και για να είμαι ειλικρινής, αυτή η έκθεση κατά τη γνώμη μου είναι περίπτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Τάιλερ ήθελε να μιλήσει. Ο κυρία Τόν Μπλουμ, καλώ ήρθατε. Φίλη της Επιτροπής. Και ο κύριος Ποτσμάτσκι από την DG Markt και τον κύριο Μπίρα από την DG Energy. Έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Ελπίζουμε να σας βολέψουμε όλους και να μιλήσετε. Σημερίζομαι τις απόψεις που ακούστηκαν, τις ανησυχίες για την έκθεση, κύριε Βίνχος. Όσον αφορά τι εκθέσει ιδίας πρωτοβουλία, εν γέννη είναι αποτελεσματικές όταν υπάρχει συνένεση ευρεία στην Επιτροπή. Αλλιώς αγνοούνται. Δεν έχουν πολιτική ισχύ. Από εσά εξαρτάται ως εισηγητής να εργαστείτε σε αυτό το πλαίσιο. Εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας δεν είναι τομείς για να κρίνεται αν κάποιες απελευθερώσεις έχουν λειτουργήσει. Θα είναι διχασμένη Επιτροπή. Πρέπει να δώσουν θέμενη αξία στη διαμόρφωση πολιτικών. Δεν θέλω να ακούγομαι εδώ σαν γυμνασιάρχης. Προσπαθώ να πετύχω το όφελος της Επιτροπής. Κατά το παρελθόν αυτό είδαμε. Είχαμε πρωτότυπες ιδέες σε εκθέσεις πρωτοβουλίες, προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε τους καταναλωτές. Και ξεκινήσαμε αυτή την έκθεση διότι περιμέναμε ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους ευάλωτους καταναλωτές της του ενεργειακού τομέα. Προσπαθήσαμε κατ' το παρελθόν σε αυτόν τον τομέα μαζί με την Επιτροπή Βιομηχανίας και την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Είναι γενικότερα θέματα που αφορούν τους καταναλωτές με αυτές τις υπηρεσίες. Κάθε τομέας έχει ιδιαιτερότητες. Μία ώρα κουβεντιάζαμε για τις επικοινωνίες και μπαίνοντας στις λεπτομέρειες. Είναι πολύ μεγάλο το πρόγραμμά μας για τα θέματα καταναλωτών στον τομέα των επικοινωνιών. Και θα περίτευε οδήποτε σχόλιο σε αυτή την έκθεση. Δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία αν αναφερθούμε στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε αυτή την έκθεση. Διότι καλύπτουμε, στο, στην προηγούμενη έκθεση καλύπτουν λεπτομέρειες. Λοιπόν, ενέργεια και ταχυδρομικές υπηρεσίες είναι αυτά που μας αφορούν, όπου δεν έχουμε άμεση ευθύνη, αλλά μπορούμε να σχολιάσουμε επικοδομητικά, τομεακά ζητήματα. Αλλαγή, διαφάνεια τιμών, συγκρισιμότητα τιμών, θέματα καταναλωτών στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Έχουμε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παράδοση πακέτων, για την ε, παράδοση της υπηρεσίας παράδοσης δεμάτων. Εργαζόμαστε και την ψηφιακή ενιαία αγορά που είναι κάτι που αλλάζει εντελώς τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Άρα από ταχυδρομικές υπηρεσίες γραμμάτων κινούμεθα περισσότερο προς τις παραδόσεις μικρών πακέτων και μεγαλύτερων δεμάτων. Εμείς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε προστιθέμενη αξία. Δεν μας πιέζει ο χρόνος, δεν είναι νομοθετικού περιεχομένου έκθεση. Θα προτιμούσα εσείς και οι σκιώδεις, εμού συμπεριλαμβανομένου, να εστιαστούμε σε ιδέες και θέμενη αξία σε βασικούς τομείς. Θέλουμε συνένεση μεγάλη για να έχουν ισχύσει στάσεις και να επηρεάσουν την καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Έτσι τα βλέπω εγώ τα πράγματα ως κοιόδης και πρόεδρος. Αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία θα ήθελα να κινηθεί η έκθεση. Η κυρία Στάιλερ. Νομίζω ότι το θέμα τα λιανικού εμπορίου της ενέργειας είναι σημαντικό και είναι στο πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σημαντικό για το πώς αντιμετωπίζονται οι καταναλωτές. Αντιμετωπίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόβλημα κόστους διαβίωσης. Έχουμε και άσπρετα Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επηρεάζουν και άλλα συναφή θέματα που αφορούν και το περιβάλλον το γενικότερο. Άρα συζητώντας τον τομέα λιανικού εμπορίου της ενέργειας να καλύπτονται οι πτυχές των καταναλωτών, διότι οι εκλογείς μας προβληματίζονται για το κόστος διαβίωσης. Πολλοί κόσμος, πολλές ενεργειακές εταιρείες συμπεριβαίνονται όπως οι τράπεζες πριν. Και οι καταναλωτές εκτίθενται σε υψηλότερες τιμές κάτι που πλήττει το εισόδημα των οικοκυριών. Οι συζητήσεις για το κόστος της ενέργειας για τους πολίτες μας είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Είναι και θέμα κρατών μελών, είναι και θέμα επικουρικότητας, αλλά να μην το λάβουμε υπόψη καθόλου όταν ο τομέας του λιανικού εμπορίου ε, ενέργειας εντάσσεται στο πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάτι που θα πρέπει να το εξετάσουμε. Το κόστος των ενέργειες καταναλωτές, όπως είπαν και άλλοι, είναι κάτι που αφορά τους εκλογείς μας. Θέλουν οι εκλογείς μας να το συζητήσουμε. Είναι πρόβλημα για αυτούς το κόστος διαβίωσης. Πρέπει να τα κουβεντιάσουμε αυτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο όταν άκουσα ότι είναι περιττή η έκθεση. Μα πώς υπάρχουν πάνω από 150 τροπολογίες, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν νομίζω ότι είναι περιττή μια έκθεση που συγκεντρώνει 150 τροπολογίες. Πρέπει να συζητηθεί. Πολλές φορές συζητήσαμε όντως και πάντα λέγαμε ότι διάφοροι τομείς πρέπει διαφορετικά να αντιμετωπίζονται. Αλλά πάντα Στιάζαμε το ενδιαφέρον μας σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα, θυμάμαι, δηλαδή τη δυνατότητα καταγγελίας σύμβασης από την πλευρά του καταναλωτή. Και σε όλες τις χώρες ε, είδαμε ότι πολλοί πάροχοι δημιουργούν δυσκολίες και δεν μπορεί να ε, γίνει καταγγελία Τώρα στη Γερμανία έχουν βελτιωθεί λίγο τα πράγματα μετά από πολλές καταγγελίες, αλλά εξακολουθούν να είναι πολλοί οι πολίτες που έχουν την εντύπωση ότι ε, καταγγελία της σύμβασης γίνεται από αυτούς μόνο μετά από τεράστιες δυσκολίες. Αυτό ισχύει για πολλούς τομείς, όχι για έναν μόνο. Αυτό όντως είναι ένα θέμα που αφορά τους καταναλωτές και πρέπει να το θεωρήσουμε πολύ σημαντικό. Άρα και μόνο εξ αυτού θεωρώ ότι δεν είναι περιττή η έκθεση. Ναι, ε, να, του προσθέσουμε αξία. Ας ακούσουμε και την Κομισιόν τώρα, στον υπόλοιπο χρόνο, για την ενέργεια ο κύριος Μπίρερ να αρχίσει και αν θέλουν και άλλοι συνάδελφοι από εκεί, για Τόν, Τόνμπλουμ ίσως και ο κύριος Ποτσμάσκι. Λοιπόν, ο κύριος Μπίρερ την, να μας ενημερώσει για τα ενεργειακά την προτινόμενη ανακοίνωση για τους ευάλωτους καταναλωτές στο τομέα της ενέργειας. Εμείς προχωράμε όχι με συγκεκριμένη ανακοίνωση για τους ευάλωτους καταναλωτές, αλλά έχουμε εκδώσει ως αποτέλεσμα της ομάδας εργασίας για τους ευάλωτους καταναλωτές σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, καταναλωτικές οργανώσεις, άλλους εμπλεκομένους. Μιλήσαμε για ορθές πρακτικές και συστάσεις και επίσης θα εκδώσουμε ανακοίνωση πιο συγκεκριμένη που θα αφορά περισσότερο το θέμα των τιμών γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό και ανησυχεί τους καταναλωτές. Θα έχουμε ανακοίνωση και ένα, για, το, για τις τιμές ε, και το κόστος της ενέργειας, ε, δηλαδή θα έχει στοιχεία για την ε, επίπτωση στους καταναλωτές. Είναι πολύ ετερογενής, διαφοροποιημένη εικόνα στα κράτη-μέλη. Και εκεί θα γίνουν ενδεχομένως συζητήσεις για ανάληψη περαιτέρω πολιτικών μέτρων. Συνεχίζουμε επίσης την εργασία μας με το κλάδο της Λιανικής, που μάλλον αργότερα θα το επεξεργαστούμε κατά τη διάρκεια του έτους και εδώ μιλάμε για θέματα καταναλωτών και αγορές λιανικής. Για την έκθεση για την ενέργεια που βλέπουμε εδώ θα βοηθούσε αυτό να το απευθύνουμε, να αναφέρεται στην έκθεση ότι αφορά τον τομέα της ενέργειας όπου έχουμε ε, ήδη εφαρμόσει μέτρα προστασίας των καταναλωτών στο τρίτο πακέτο ενέργειας όπου μιλάμε για διαφάνεια τιμών, δικαίωμα αλλαγή παρόχου, προθεσμίες για την αλλαγή παρόχου, διάφορα ε, θέματα που πρέπει να εφαρμοστούν από τα κράτη-μέλη ή από κράτη-μέλη που κάναμε έλεγχο και τώρα ε, επιβάλλουμε αυτά τα, εφαρμόζουμε αυτά τα μέτρα. Και για τους ευάλωτους καταναλωτές, τα κράτη-μέλη θα πρέπει οπωσδήποτε να ορίσουν τις ευάλωτες κατηγορίες και θα το δούμε αυτό αν έχει γίνει. Επίσης συστήνω με προσοχή για τον ενεργειακό τομέα ε, σχετικά με το αίτημα των ευάλωτων καταναλωτών, των ευάλωτων οικονομικά ε, καταναλωτών που θα πρέπει να ωφελούνται από την μείωση των τιμών ενέργειας. Αυτό το μονοπάτι το ακολούθησαν αρκετά κράτη-μέλη, αλλά η εφαρμογή είναι θέμα επικουρικότητας, γιατί σε άλλα κράτη-μέλη τους δίνουν οικονομική υποστήριξη, κάποιο επίδομα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους. Και αυτός είναι νόμιμος και θεμητός τρόπος και αποτελεσματικός επίσης. Εμείς το έχουμε συζητήσει στην ομάδα εργασίας για τους ευάλωτους καταναλωτές και το έχουμε δεχτεί αυτό το μέτρο. Μπορείτε να μας πείτε τι τεκμηρίωση υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμη και πότε θα ε, έχουμε την ε, ανακοίνωσή σας η μελλοντική ανακοίνωση για το κόστος και τις τιμές ε, θα είναι διαθέσιμη πολύ σύντομα. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος για το ε, ακριβές χρονοδιάγραμμα. Τις επόμενες εβδομάδες ή σε ένα μήνα. Έχουμε κάποιες πληροφορίες ε, για τις βέλτιστες πρακτικές ε, και την υποστήριξη των ευάλωτων καταναλωτών που τις έχουμε διαθέσει στον ιστότοπό μας, ε, στην ομάδα εργασίας για τους ευάλωτους καταναλωτές. Έχουμε κάποιες συστάσεις εκεί. Νομίζω ότι αυτά είναι τα σημεία μεγάλου ενδιαφέροντος. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τον τομέα της προστασίας καταναλωτών. Υπάρχει, υπάρχουν και κάποια στοιχεία στο νησότοπό μας σχετικά με τους ευφυείς μετρητές στα νοικοκυριά και το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι ισχυρισμοί οι οποίοι δεν, ε, ε, ε, δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί. Γι' αυτό εμείς ενθαρρύνουμε την ανάλυση κόστους κόστους-οφέλους στα κράτη-μέλη σε σχέση με το, τους ευφυείς μετρητές. Γιατί θέλουμε να τους προωθήσουμε σε ένα πλαίσιο που πραγματικά θα είναι επωφελές για τους καταναλωτές. Ναι, πράγματι, αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Κύριε Τούνμπεργκ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους ε, αξιότιμους ευρωβουλευτές ε, για την, ε, το συμβιβαστικό τους πνεύμα. Περιμένουμε αγωνίως την επόμενη εκδοχή του κειμένου και συμφωνούμε με την άποψη ότι δεν είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για επιπλέον νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύτερα είναι να εφαρμόσουμε και να ε, τροποποιήσουμε τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναλυφθεί και δρομολογηθεί. Τούτων λεχθέντων, οι τροπολογίες ε, και αυτά τα οποία είπατε είναι πάρα πολύ χρήσιμα για την τελειοποίηση της ε, έκθεσης, όπως επίσης και την οριοθέτηση των διαφόρων επιπέδων ευθύνης γιατί μερικά κάποια ευθύνη επαφίεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποια ε, ευθύνη, κάποιο τμήμα της ευθύνης στα κράτη-μέλη δεν είναι απολύτως σαφή τα πράγματα. Οι κατατεθείς τροπολογίες ε, δείχνουν ότι ε, το όφελος των καταναλωτών έχει ήδη ενσωματωθεί ε, στην νομοθεσία για το μίσο όπως οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η ενέργεια, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και μάλιστα θεωρούν ότι είναι, θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητες στο πλαίσιο του θεματολογίου που αφορά τους καταναλωτές ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση για τους καταναλωτές. Γνωρίζουμε πόσο περίπλοκο περίπλοκη και δύσκολη είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζει ο κάθε καταναλωτής. Η οδηγία προστασίας καταναλωτών και η έναρξη ισχύω της θα βοηθήσει επίσης. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας και τον εναλλακτικό ε, και τον ε, ε, ηλεκτρονικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών που θα βοηθήσει πολύ ειδικότερα στις χώρες που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ως συνήθις προσέγγιση για την επίλυση των διαφορών. Νομίζω επίσης ε, και τώρα αυτό είναι πρακτική ενημέρωση, η αξιοπιστία των εργαλείων ε, σύγκρισης είναι πάρα πολύ σημαντική για ε, τους τομείς αυτούς. Είναι πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές ως εργαλείο και γι' αυτό Έχουμε συχνά διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους εθνικούς ρυθμιστές, τους καταναλωτές, τους επιχειρηματίες. Έχουμε, εκπονούμε και μια μελέτη, τον Ιούλιο του 2014 θα δημοσιευθεί, για να έχουμε μια ευρύτερη εικόνα της αξίας των εργαλείων αυτών ε, και του ωφέλους τους για τους καταναλωτές και το τι δεν δουλεύει καλά βέβαια. Όσον αφορά τις τροπολογίες που έχουν να κάνουν με τις οργανώσεις τις καταναλωτών, θα ήθελα να τονίσω ότι η χρηματοδότηση των εθνικών οργανισμών παραμένει ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων ή των εθνικών ε, αρχών. Εμείς ευρωπαϊκό, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, χρηματοδοτούμε ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Είναι σημαντικό για μας αλλά προσπαθούμε ενεργά να πείσουμε τις εθνικές αρχές και τις κυβερνήσεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε εθνικό επίπεδο. Όσον αφορά τώρα τους ευάλωτους καταναλωτές, ε, Υπάρχει και έκθεση από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση, αλλά και εμείς το παίρνουμε πολύ σοβαρά αυτό το, θέμα, το θέμα, οπότε και εμείς εκπονούμε μία ευρεία μελέτη που εστιάζει και στην ενέργεια αλλά και σε άλλους τομείς και σε, άλλες, σε άλλους τομείς που έχουν αρχίσει πρόσφατα να αναπτύσσονται και προσπαθούμε να δούμε τα, τις τάσεις ευαλωτότητας. Ελπίζουμε να είναι διαθέσιμη η έρευνα το 2015 για να μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη θεώρηση του θέματος και να το αντιμετωπίσουμε διεξοδικά. Ε, ο συνάδελφος από τη Γενική Διεύθυνση ε, ενέργειας ε, συνεργάζεται πολύ μαζί μας. Έχουμε ομάδες εργασίας ε, στις οποίες ε, συμμετέχουν πολύ ενδιαφερόμενοι φορείς, ρυθμιστές από τα κράτη-μέλη. Όλοι συμμετέχουν και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις και όλοι δουλεύουμε για την παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών. Η επικουρικότητα γίνεται σεβαστή στους διάφορους τομείς, αλλά σημαίνει επίσης ότι είναι και η ανάπτυξη, η εξέλιξη διαφορετική σε διάφορα κράτη-μέλη και μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς μπορούν να επιληθούν προβλήματα. Για την έκθεση, για την ευαλωτότητα, ε, έχουμε ε, μελέτες και για τη διαχείριση των ε, δεδομένων και συνεχίζουμε για την ε, συλλογική μετάβαση, για ε, τις κοινέ αγορές και ελπίζουμε να ε, μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε τις σχετικές μελέτες την επόμενη χρονιά. Υπήρξαν κάποιες τροπολογίες για τις οποίες η Γενική Διεύθυνση, οι άλλες γενικές ευθύνσεις έχουν πολύ συγκεκριμένα σχόλια να κάνουν. Έχετε ένα-δύο λεπτά στη διάθεσή σας. Γρήγορα θα σας τα πω πρώτα απ' όλα γιατί είναι τα γενέθλιά μου και δεύτερον πρέπει να φύγω. Λοιπόν, δεν θα πω σε τροπολογίες. Ε, νομίζω πάντως ότι πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Δύο παρατηρήσεις παρόλα αυτά. Πρώτον, ε, εκδώσαμε τον Δεκέμβριο έναν οδικό ε, χάρτη για τα διασυνοριακά ζητήματα, τα πακέτα, την τιμολόγηση. Ε, και υπάρχουν πολλές δράσεις που έχουν δολοπολογηθεί αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά την έκθεση εφαρμογής, η οποία λογικά θα δημοσιευθεί μέχρι την επόμενη φορά που θα ε, έρθουμε εδώ, είναι προνόμιο της επόμενης επιτροπής να το παρουσιάσει, γιατί θα έχει περισσότερο χρόνο να το επεξεργαστεί. Οπότε πιστεύω ότι σε, σε ένα χρόνο περίπου θα έχουμε τα αποτελέσματα. Μία τελική παρατήρηση για την 143 τροπολογία Χαίρομαι που υπάρχει καλύτερη επισκόπηση των ε, διαδικασιών καταγγελιών και στα κράτη-μέλη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως το άρθρο 19 της ε, οδηγίας δεν το προβλέπει αυτό. Θα πρέπει να αλλάξουμε την ομοθεσία επ' αυτού. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα επικουρικότητας και υπάρχει και θέμα πόρων. Όπως καταλαβαίνετε πρέπει να ε, κάνουμε περικοπές 5% στην Επιτροπή, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το διοικητικό άχθος είναι διόλου αμεληταίο. Ουσιαστικά θα υπάρχει ένας υπερρυθμιστής στην, ε, στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Εγώ θα μπορούσα να είμαι υπέρ αυτού, γιατί αυτό θα σήμαινε περισσότερες ε, ε, θέσεις εργασίας, ίσως και περισσότερα καθήκοντα για μένα τον ίδιο, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε τις συνέπειες και πρέπει να σας προειδοποιήσω. Όταν συζητήσετε λοιπόν αυτές τις τροπολογίες, παρακαλώ λάβετε υπόψη όλες τις προεκτάσεις ε, ή δώστε μας ε, περισσότερους ε, πόρους για να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή... Κα... χρόνια πολλά ήθελα να σας ευχηθώ εφόσον είναι τα γενέθλιά σας. Λίγο σύντομα συνάδελφοι γιατί πρέπει να φύγουν και οι διερμηνείς. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια έκθεσή σας ε, για τις 11 Φεβρουαρίου. Ε, ίσως θα έχετε χρόνο να, να συζητήσετε και με τους σκιώδεις για να το συζητήσετε περισσότερο. Αν θέλετε λίγο περισσότερη περίοδο προβληματισμού μπορώ να σας δώσω, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει πίεση χρόνος προς την έκθεσή σας. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Ε, θέλω να ευχαριστήσω όλους για την κριτική σας για τα θετικά σας σχόλια. Συνοψίζοντας, λέω μόνο ότι μετά τη συζήτηση είναι σαφές ότι δεν θέλουμε κι άλλες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Είναι σημαντικό να δούμε τις διαφορετικές ε, εντάσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις τομεακές και οριζόντιες ε, προσεγγίσεις ε, ευχαριστώ τον πρόεδρο που αναφέρθηκε στις τηλεπικοινωνίες και συμφωνώ επίσης μαζί του ότι χρειάζεται μια ευρεία συνένεση ε, πάνω σε αυτά τα θέματα. Έχω την αίσθηση ήδη ότι υπάρχει μια βασική ιδέα που θεωρεί σημαντική και απαραίτητη την έκθεση και χρήσιμη και τις προτάσεις που άκουσα θα προσπαθήσω να τις επεξεργαστώ και να επανέλθω και στην πρόταση του Προέδρου μας. Ευχαριστώ πολύ και να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά στο συνάδελφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωραία, σας ευχαριστούμε όλους πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Βάιντεν Χόλτσερ για την επικοδομητική του απάντηση. Στις 3 ξανά που θα έχουμε τον Υπουργό κύριο Χατζηδάκη, πρώην Ευρωβουλευτή και συνάδελφό μας. Φαντάζομαι ότι πολλοί θα ενδιαφέρονται για το τι έχει να μας πει για την ελληνική Προεδρία. Ε, θα αρχίσουμε ακριβώς στις 3. Ευχαριστώ.